Good Ας ξεκινήσουμε, παρόλο που δεν είναι πολλοί παρόντες. Έχει περάσει ήδη ένα τέταρτο. Ας ξεκινήσουμε με τα επόμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης. 7. Την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ειδικής Τράπεζας, στο σημείο 7. Στην κυρία Μαρίζα Ματίας δίνω το λόγο, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας για τη συνεργασία των με τους συναδέλφους, συναδέλφους των διαφορετικών ομάδων που τις τελευταίες ημέρες είχαμε διμερείς συναντήσεις και προχωρήσαμε κάπως τη δουλειά για τις συμβιβαστικές τροπολογίες σε σχέση με την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δώσω μια σύντομη υπεξήγηση, αυτό που προσπάθησα να κάνω στις ε, συμβαστικές προτάσεις τροπολογίας που διανεμήθηκαν και συζητήθηκαν, είναι αφενός <clears throat> να εκπονήσω κοινέ προτάσεις τροπολογίας, πάντα όπου αυτό ήταν δυνατό να γίνει, και σε άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη απόκληση τοποθετήσεων, προσπάθησα να δραχθώ της ευκαιρία. με θετικό πνεύμα από πλευράς των προτάσεων κάποιων συναδέφων για τη διατύπωση των προτάσεων ώστε να έχουμε μια νέα βάση με αυτή την αναδιατύπωση για τη διαπραγμάτευση και για τη συνεννόηση. Αυτή ήταν η στρατηγική που ακολουθήθηκε λοιπόν. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία κατέθεσα ήδη στους διάφορους 24 συμβαστικές τροπολογίες στους συναδέλφους ιδιαίτερα σε σχέση με τις παραγράφους που αρχικά ε, εντασσόντουσαν σε σχέση με τις προτάσεις και συμβιβασμούς που θέλουν πολλούς τομείς να καλύψουν όπου υπάρχουν διάφορες ιδέες και τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και που πιστεύω ότι μπορούμε έτσι να καταφέρουμε, καταφέρουμε καταφέραμε να βρούμε μια διατύπωση που μπορεί να μας είναι χρήσιμη και ικανοποιητική για όλους και μπορούμε να τη συμμεριστούμε όλοι και που αφορούν θέματα διαφορετικά αυτά για τη διαφάνεια, θέματα τα οποία συσχετίζονται με το SMP τις δράσεις αυτές, ένα κοινό ολόκληρο θέμα πλαίσιο για τροπολογίες που κατατέθηκαν και που προσπάθησα να δώσω συνέχεια με συμβαστικές τροπολογίες σε αυτές. Αυτό που θα κάνω είναι κάποια γενικά σχόλια. Δεν θα εξηγήσω τα σχετικά με κάθε μία τροπολογία. Δεν έχει νόημα αυτό σε αυτό το πλαίσιο. Πολύ συνοπτικά λοιπόν θα ήθελα να επεξηγήσω κάποια πράγματα και να δώσω κάποια σχόλια για τις προτάσεις που έχουμε στο τραπέζι τώρα, ώστε μετά να ακούσω τα σχόλια από τους συναδέλφους και να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και να προχωρήσουμε λίγο στη συζήτηση πρώτα. Το πρώτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω αφορά το γεγονός ότι εγώ συνεχίζω να κατανοώ ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ κάτι, να υπογραμμίσουμε το πλαίσιο της νομισματικής ε, ε, πολιτικής, την εφαρμογή αυτής της νομισματικής πολιτικής. Γιατί πρέπει να βρούμε ένα τέτοιο πλαίσιο που μπορούμε όλοι να το ε, δούμε από κοινού όταν έχουμε χαμηλό ποσοστό ανάπτυξης, έχουμε προβλήματα σε σχέση με πιστώσεις και δάνεια και έλλειψη δυναμικής για τα δάνεια και τις πιστώσεις το που επιβαρύνει την κατάσταση και που αυτό το οποίο συνέβη σε σχέση με το ε, εξάμεινο αυτό και για την πρόταση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη δική μου πρόταση, συμμεριζόμαστε όλοι αυτή την άποψη νομίζω. Έχει τεράστια σημασία η οικονομική ανάπτυξη λοιπόν. Τεράστια σημασία. Και είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη αυτό το θέμα της ανάπτυξης και να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα. Το δεύτερο ζήτημα αφορά το θέμα των όρων και προϋποθέσεων και τους περιορισμούς για τις τράπεζες. Και εδώ πάλι έχουμε κάποιες προτάσεις και μπορούμε να συμμεριστούμε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για τα κράτη, που αν υπάρχουν για τα κράτη πρέπει να υπάρχουν και για τις τράπεζες εξίσου. Είναι προφανές, είναι πρόδειλο αυτό. Και πολλές από τις προτάσεις ε, που κατατέθηκαν και αυτοί που καταθέτω ασχολούνται με το ότι θεωρούμε εμείς ότι αυτές οι μεταφορές κονδυλίων πρέπει να συνεισφέρουν για την αύξηση των πιστώσεων στην οικονομία, ιδιαίτερα αύξηση πιστώσεων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτά για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί χωρίς αυτή την δέσμευση όλη η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής αμφισβητείται, υπονομεύεται. Διάφορες συζητήσεις ε, που έγιναν, εγώ θα αναφέρω τα εξή. Πρώτα απ' όλα και αυτό αφορά το, τους όρους υπό τους οποίους θα διεξαχθεί η νομισματική πολιτική και η αποτελεσματικότητα που θα έχει αυτή για τις συζητήσεις κάποιων από τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους συναδέλφους σε σχέση με τα μη συμβατικά μέτρα, την αποτελεσματικότητα και κάποιους μη κάποια μη επιθυμητά αποτελέσματα που μπορεί να παρουσιαστούν. Θεωρώ ότι πρέπει εδώ να επισημάνουμε τη σημασία που έχει, που θα μπορεί να έχει η δυνατότητα του να διευκολύνουμε ένα quality mix, ένα policy mix, ένα μείγμα πολιτικών για την νομισματική πολιτική και μια δημοσιονομική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι θέματα αυτά που πρέπει να τα συζητήσουμε πιστεύω σε αυτή την έκθεση. Σε κάποιες τροπολογίες, αρκετές τροπολογίες από αυτέ που κατατέθηκαν, εμφανίστηκαν ανησυχίες που συσχετίζονται με τις ε, επιπτώσεις ε, που θα έχουν αυτά όλα σε σχέση με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι τροπολογίες που καταθέτω είναι να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για τους διαφορετικούς τύπους ενεργητικού κεφαλαίου για να έχουμε το επίπεδο έκθεσης και τη χρήση αυτών των κεφαλαίων και τη δυνατότητα που μπορεί να ε, τύχουν, των δυνατοτήτων που μπορεί να τύχουν αυτές οι δράσεις. Από την άλλη πλευρά, στην έκθεση για συμβαστικές τροπολογίες που καταθέτω, αναζητώ να εκφράσω κάτι αυτό τι είναι. Το μέλημα, η ανησυχία και αυτό εκφράστηκε και από διάφορους ε, συναδέλφους πέρα από μένα για τις μη ισόρροπες ε, σχέσεις που υφίστανται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι ανισότητες είναι συνέπεια ροών κεφαλαίων και γνωρίζουμε επίσης ότι μπορούν να διαμφισβητήσουν, να υπονομεύσουν ε, την ενότητα και τη συνοχή του ευρώ. Είναι ένα από τα θέματα που αναζήτησα να αντιμετωπίσω και είναι αυτό κάτι το οποίο αφορά και ανησυχίες των συναδέλφων. Πέρα από όλα αυτά τώρα, το σύνολο των τροπολογιών σχεδιάζουν μία διέξοδο, καταδεικνύουν μία διέξοδο σε σχέση με την νομισματική πολιτική και τα προβλήματα όσον αφορά το 2011, σε σχέση με τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και την εντολή που θα έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι μία συζήτηση που συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Θέλω σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες αυτή την αξιολόγηση να κάνουμε σε σχέση με την νομισματική πολιτική μέσα στο πλαίσιο της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εξουσιών της, των αρμοδιοτήτων της. Μέσα σε αυτή την πρώτη αντιμετώπιση, σε αυτή την πρώτη φάση, παρόλα αυτά πιστεύω ότι δεν πρέπει να αποκλείσουμε ούτε τη συζήτηση, ούτε την εξέταση για τους στόχους της νομισματικής πολιτικής και σε σχέση με τον στόχο της καταπολέμησης του πληθωρισμού να έχουμε την εντολή αυτή για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα συμμετέχει στην εξέταση αυτή αλλά να συζητήσουμε και τα άλλα συναφή θέματα. Επίσης, σε σχέση με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα προγράμματα προσαρμογής και λιτότητας και την εκπόνηση μέτρων για τη διαθροτική πολιτική από την νομισματική πολιτική, σε σχέση με τα θέματα εντολής ε, που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά τα δύο θεματικά πλέγματα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη στη συζήτηση. Για να ολοκληρήσω και δεν θα εμβαθύνω σε όλα τα θέματα που μας απασχόλησαν, σε δεύτερο γύρο θα καλύψω άλλα περισσότερα θέματα. Σε αυτή την πρώτη φάση θέλω να πω καθώς είχαμε πολλές τροπολογίες από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες ότι πρέπει να υπάρχει ενίσχυση διάχυσης, διάδοσης πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πρακτικά συνεδριάσεων, ε, στοιχεία όσον αφορά τα, ε, το ενεργητικό και άλλα συναφή θέματα η δική μου, ο δικός μου προσανατολισμός στις ε, τροπολογίες που καταθέτω ως συμβασικές τροπολογίες ήταν το πνεύμα αυτών των τροπολογιών προσπαθεί να βρει τις προτάσεις, να εντάξει τις τροπολογίες που κατατέθηκαν σε ένα πλαίσιο για ευρύτερη συνένεση και διαφάνεια, για μεγαλύτερη διαφάνεια. Νομίζω επ' αυτού μπορούμε να συμφωνήσουμε, συμφωνούμε και μπορούμε να συνεχίσουμε στην εμβάθυνση αυτών των θεμάτων. Αναμένω να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και θα επανέλθουμε μετά με αυτή τη συζήτηση συζήτηση θα δώσουμε συνέχεια. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ματίας. Δεν υπάρχει μέλος, μέλος του ΕΛΚ να πάρει το λόγο, οπότε δίνω σοσιαλιστές το λόγο. Και στο τέλος της συζήτησης, αν, δεν, αν υπάρχει κάποιος του ΕΛΚ, θα του δώσω το λόγο. Για τους σοσιαλιστές, ο κύριος Άνιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά από την τελευταία συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή είχαμε καρποφόρα συνεργασία με τον εισηγητή και με τη συγγήτρια και του Σκιώδης. Ήρθε σε επαφή η κυρία Ματίας με όλους μας για να καταλήξω συμβιβασμό για την έκθεση που για το Κοινοβούλιο είναι μια ευκαιρία να γνωμοδοτήσουμε όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κυρίως την μακροοικονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Να υπενθυμίσω ότι η έκθεση της Μάριαν Τίσεν που εν μέρη ασχολείται με θέματα που αναφέρονται και στην έκθεση Ματίας όπως τον έλεγχο της Τρόικα ε, συνεκέρασε ε, πολλέ απόψει στην Ολομέλεια και συγκέντρωσε την υποψηφία στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα. Έχω πεποίθηση στη συλλογική μα ικανότητα να κατορθώσουμε συγκεντρώσουμε μεγάλη πλειοψηφία ε, όσον αφορά την έκθεση τη κυρία Ματία. Έτσι δε περαιτέρω, διότι οι σημαστικές προτάσεις που μας κάνει η συγγήτρια αντιπροσωπεύουν μια σημαντική προσπάθεια την οποία θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Θα ήθελα να τη συγχαρώ και για τη μέθοδο εργασία που ακολούθησε αλλά και για το περιεχόμενο των προτάσεών της που θεωρώ ότι εγκατοπτρίζουν καλά τις απόψεις των διαφόρων ομάδων. Η ανάλυση της νομισματικής πολιτικής που παρουσιάζει τις προτάσεις της είναι κάτι ιδιαίτερα ισορροπημένο και η γλώσσα που χρησιμοποιεί δείχνει πόσο περίπλοκη είναι η μακροοικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης. Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέσα, όπως το, ε, τα δύο που αναφέρει, καθώς και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τις περιφερειακές χώρες όπως αποκαλούνται, που είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό, θεωρώ ότι οι προτάσεις εκεί της εισηγήτριας αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής μας. Τέλος, οι προτάσεις της απηχούν τις θέσεις που ασπίστηκε το Κοινοβούλιο στον αφορά το θέμα αυτό, δηλαδή το Ταμείο της Διάσωσης που είναι κάτι αγαπητός φιλελευθέρους ή ε, την δυνατότητα τη δημοσιονομική την αντικυκλική ε, που υπερασπίζεται η ομάδα S&D και αυτό είναι αξιέπαινο. Ε, για να κλείσω αγαπητοί συνάδελφοι δεν μπορώ παρά να σας ενθαρρύνω να μελετήσετε τις προτάσεις της εισηγήτριας με νέο πνεύμα, χωρίς προκαταλήψεις. Νομίζω ότι θα βρείτε ότι είναι ικανοποιητικά αυτά που αναφέρονται, όπως και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χωανιόκ. για την Άλτε έχει το λόγο και ο Στεμόσα. Ευχαριστώ πολύ, Παύλο. Μια και σήμερα είσαι εσύ πρόεδρος, θα μιλήσω ισπανικά. Και έτσι, σαν πρώτη φορά, ως σηματοδότηση ε, φιλικής σχέσης ε, και θετικής ατμόσφαιρας. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή την έκθεση, μια και είχαμε μια πολύ γόνιμη συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο όπου δεν είχαμε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες και από την φιλελεύθερη ομάδα φοβόμαστε κάπως ότι δεν θα υπήρχε ένα κοινό σημείο, ένα κοινό σώμα από το οποίο θα μπορούσαμε να πετύχουμε μεγαλύτερες συνενετικές θέσεις από το σώμα. Βλέπουμε στιγμές ε, μεγάλων προβλημάτων και ναυαγίων στις αγορές και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η συζήτηση αυτή μαγνητίζει την προσοχή όλων των μέσων και υπό αυτό το πρίσμα υπήρχαν ανησυχίε στην ομάδα μου. Αλλά δεδομένων τώρα αυτών των πρώτων τροπολογιών, συμβιβαστικών τροπολογιών, σε αυτή την πρώτη φάση όπως κατατέθηκαν, εγώ προσωπικά χωρίς να γνωρίζω ακόμα την άποψη των συναδέφων είμαι ικανοποιημένο μπορώ να πω. Μια και είδα μια προσπάθεια που έγινε για να προσπαθήσει να εντάξει τροπολογίες διαφόρων ομάδων στις διάφορες συμβιβαστικέ τροπολογίες που κατατέθηκαν. Μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο, γρήγορα θα αναφερθώ λέγοντας ότι συμφωνούμε με τις τροπολογίες 2, 4, Προσωπικά κάνω λόγο για αυτή την περίπτωση, για την 2 και την 4, την 9, την 10, την 12, 14, 15, 17, 18, 19, 16, 18, 19, με συγχωρείτε, 20, 21, 22, 24. <clears throat> για τις άλλες τροπολογίες θα, έχουμε, θα είχαμε κάποιες αμφιβολίες. Μπορούμε να δούμε και να εξετάσουμε κάποιες εναλλακτικέ διατυπώσεις. Αλλά καταρχήν θεωρούμε ότι είναι καλό ένα μέρος του έργου που έχει επιτελεστεί με αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες και όταν στο τέλος θα έχουμε περισσότερες και άλλες ιδέες για τις συμβαστικές τροπολογίες πάλι μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια για να εντάξουμε και τροπολογίε άλλων ομάδων και ιδιαίτερα σε σχέση και με τι δικέ μα θέσει φιλελεύθερης, ε, φιλελεύθερης ομάδας ε, για το Target 2, για τους, ε, τα θέματα που συνάπτονται του Target 2 για τις, με, αυτές τις, με αυτή την προσδοκία ελπίζουμε θα έχουμε περισσότερες συναντήσεις για να καταλήξουμε σε ένα σκαρίφημα αυτής της έκθεσης που μπορεί να γίνει αποδεκτό να υπερψηφιστεί από όλους. Πολλές τροπολογίες φυσικά θα πρέπει στο τέλος να ψηφιστούν και κάθε ένας θα πρέπει να διατηρήσει και τη δική του θέση και να καταθέσει τις δικές του τροπολογίες. Αλλά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και θα πρέπει να είμαστε ικανοί να βρούμε κοινέ θέσει. Δεν θα εξυπηρετούσαμε την, ε, τα συμφέροντά μα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν κατακαιρματιζόμαστε και δεν είχαμε κοινέ θέσει. Υπάρχουν κάποιε ε, ε κόκκινε γραμμέ, ε, διαχωριστικέ γραμμέ όσον αφορά την φιλελεύθερη ομάδα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια κόκκινη γραμμή ότι η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα μπορούσε να διαμφισβητηθεί. Για μας αυτό είναι απειρόβλητο, είναι στο απειρόβλητο. Είναι χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η αυτονομία της και η ανεξαρτησία της. Και πιστεύουμε ότι η ζώνη ευρώ δεν είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Το ευρώ δεν είναι το δολάριο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και σε σχέση με τις ε, επεκτατικές πολιτικές που ακολουθούν σε σχέση με Άλλος η δική μου ομάδα λέει ότι η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι το μεγάλο κεκτημένο, η μεγάλη αξιοπιστία, το μεγάλο θετικό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή της. Όταν αμφισβητείται αυτό όπως σε κάποιες χώρες πρέπει να πούμε ότι το μεγάλο κεκτημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από την ενιαία εσωτερική αγορά είναι το ενιαίο νόμισμα και η αξιοπιστία το ευρώ και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και σαν σημείο πιθανών συζητήσεων λοιπόν θα πρέπει να δούμε με κριτικό πνεύμα κάποια από τα μη συμβατικά μέτρα <clears throat> όπως ε, συζητούνται και προτείνονται τους τελευταίους μήνες Μπορεί να μην συμμεριζόμαστε πάρα πολλέ ε, τροπολογίε, αλλά παρόλα αυτά για μα είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα αυτό και που μπορεί να δημιουργήσει στη συνέχεια να προκαλέσει περαιτέρω συζητήσει και αν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω συζητήσεων. Ευχαριστώ για την προσπάθεια και το θέμα των τροπολογιών αυτό έτσι όπως προχώρησε μπορεί να επιλύσει πολλά θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή τη χειρονομία που την αξιολογούμε και την εκτιμούμε ιδιαίτερα. Εξ ονόματος των Πρασίνων δεν έχουμε πάλι κανέναν εδώ. Και εξ ονόματος των FR έχουμε εσάς. Παρακαλώ έχετε τον λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. παραδοσιακός εισηγητής της ομάδας μας για τα θέματα της ΕΚΤ είναι ο κύριος Σάπινγκ, ο οποίος όμως δεν είναι παρόν σήμερα και γι' αυτό θα σας μεταφέρω συνοπτικά τις παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Ο κύριος Σάπινγκ είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από τις προτάσεις τις συμβιβαστικές τις οποίες κάνει ο εισηγητής. Η εισηγήτρια μάλλον. Η κυρία Ματίας λέει ότι καλύπτει τις τροπολογίες μας, αλλά αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Ο κύριος Σέφινγκ θεωρεί ότι περισσότερες από τις προτάσεις του θα ληφθούν υπόψη στις τελικές συμβιβαστικές ε, ε, τροπολογίες. Εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, ο εισηγητής μας θα ζητήσει, ο συντονιστής μας μάλλον, θα ζητήσει ξεχωριστή ψηφοφορία. Δεύτερον, ο κύριος Σάπινγκ προτείνει να μην υπάρχουν παραπομπές σε θέματα χρηματοδότησης ε, με νομισματικά μέσα. Ιδιαίτερα την παράγραφο 13 η οποία προβλέπει ότι θα πρέπει τα κέρδη ε, από το δημόσιο ελληνικό χρέος σαν παράδειγμα τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διανεμηθούν. Ε, εδώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην αρχική διατύπωση και στη συμφωνία στην οποία κατέληξε στις αρχές της ε, τρέχουσας εβδομάδας ε, το Eurogroup. Κανονικά τα χρήματα θα πρέπει να διανεμηθούν στις κεντρικές τράπεζες ε, ανάλογα με το ποσοστό το οποίο κατέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή είναι πολιτική απόφαση όμως. Τρίτον, ο κύριος Άπινγκ θεωρεί ότι οι τελικές, οι τελικές ευχές για επιπλέον ε, δημοσιονομικά μέσα απαράδεκτον. Αντικυκλικά ταμεία τα οποία θα γίνονται αντικείμενο διακήρυσης ε, κοινής, όπως επίσης αδειοδοτήσεις για πιστοτικές δραστηριότητες. Όλα αυτά είναι προτάσεις και θέματα τα οποία δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε δεκτά και είναι θέματα τα οποία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ΕΚΤΑΦ. Και τέταρτον, ο κύριος Τσάπεν δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη αμφισβήτησης του καθεστώτος της ΕΚΤΑΦ όπως επίσης και των στόχων της, οι, οποίες οποίοι ξεκαθαρίζονται στη συνθήκη. Θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι απαιτήσει διαφανείας και υποστηρίζει τη συμβιβαστική πρόταση για την δημοσίευση του ε, Διοικητικού Συμβουλίου, των πρακτικών μάλλον, των συνεδριάσεων ε, του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Λοιπόν, ε, κλείνοντας, η ομάδα μας δεν θα μπορέσει να υποστηρίξει την έκθεση της κυρίας Ματίας. Αυτή είναι η θέση του κυρίου Άπινγκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την αποσαφήνιση διότι ο σκιώδης εισηγητής είναι ο κύριος Έπινγκ, δεν το ανέφερα αυτό και ζητώ συγγνώμη για αυτό. Χωρίς να καθυστερούμε λοιπόν τώρα, δίνουμε τον λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ματίας. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Πολύ σας ευχαριστώ. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω για τα σχόλια που έγιναν. Υποστηρίζω τους συνάδελφους και για την υποστήριξη των συναδέλφων σε σχέση με αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες με εξαίρεση φυσικά αυτά τα οποία ακούσαμε από την ECR, από τους συντηρητικούς. Έχουμε ένα θετικό λοιπόν περιθώριο έτσι για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πλειοψηφική συμφωνία από πλευρά της Επιτροπής μας. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να υπάρξει αυτή η συμφωνία λοιπόν. Μόνο κάποια λίγα σχόλια, πολύ εξειδικευμένα, πολύ συγκεκριμένα, γιατί προφανώς δεν θα σχολιάσω όλα όσα αναφέρθηκαν. Εξάλλου ευχαριστώ αν μπορούν να αποστείλουν αυτά τα σχόλιά τους οι συνάδελφοι και γραπτός για να μπορούμε να τα εξετάσουμε καλύτερα. Θα ήταν πολύ ευπρόσδεκτο αυτό. Αλλά ακόμα και έτσι κιόλα θα ήθελα, αν γίνεται, να κάνω κάποια σχόλια πρώτα. Τώρα, σε σχέση με το σημείωμα το οποίο, ή την παρατήρηση που έγινε από πλευρά του συναδέλφου για την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η παρατήρηση αυτή. Εγώ θα ήθελα απλά μόνο να σχολιάσω και να αποσαφηνίσω κάτι και να πω ότι η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην άσκηση της εντολής της για την νομισματική πολιτική όπως γνωρίζουμε δεν αμφισβητείται από την έκθεση ή από τις τροπολογίες αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι, λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που έγιναν και τα σχόλια που έγιναν, ακριβώς να μην αμφισβητήσουμε εδώ αυτή την ανεξαρτησία, να μην την υπονομεύσουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο πλαίσιο άσκησης της εντολής του πρέπει, πρέπει να δράσει. Αλλά ένα από τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε και πρέπει να εξετάσουμε είναι θεωρώντας αυτό ως δεδομένο και εκτιμένο και ως εγγύηση για τις ε, δεσμεύσεις αυτές, το ερώτημα που θέτω είναι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ή όχι το δικαίωμα να αποφασίσει σε σχέση με τα θέματα τα οποία αφορούν την ε, έντολη αυτή. Και πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα νομίζω, διότι η αποσαφήνιση αυτή είναι αναγκαία, πρέπει να υπάρξει. Από την άλλη πλευρά διατηρούμε αυτή τη γραμμή όπως ε, αναφέρθηκε και από πλευρά συναδέλφου. Αλλά λαμβάνοντα υπόψη ότι και για μα είναι σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενεύει πέρα από το πλαίσιο τη εντολή τη πολλέ φορέ, αυτό αφορά άλλο σχόλιο το οποίο έγινε, κυρίω όσον αφορά την παρέμβαση για τα προγράμματα προσαρμογής. Έχει παρέμβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα σε αυτό το πεδίο και γι' αυτό αν παραμένει ανοιχτό αυτό το θέμα θα έλεγα και πρέπει να το εξετάσουμε. Αυτό συσχετίζεται επίσης και με αυτό που αναφέρθηκε από τον συνάδελφο της ECR, της κοινοβουλευτικής ομάδας ECR, σε σχέση με μια άλλη ε, συμβαστική τροπολογία που είπε ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει λέει αποδεκτή. Λοιπόν αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να λάβουμε υπόψη σε σχέση με αυτά τα θέματα τούτο το ότι η αναπροσαρμογή, η αναδιάρθρωση, η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι κατά κάποιο τρόπο η προσπάθεια να αποφευθεί να έχει κέρδος κέρδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από αυτή την κατάσταση. Αυτό το αναγνωρίζει και η ίδια η έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι τίποτα καινούριο αυτό το οποίο αναφέρουμε και γι' αυτό όταν έχει περισσότερα τέτοια έσοδα από τέτοιου είδους κέρδη θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Αυτά τα κέρδη στη συνέχεια διανέμονται και θέλουμε να δούμε η μεταφορά αυτή, η χρηματοοικονομική μεταφορά σε σχέση με την Ελλάδα πώς θα μπορεί να ε, γίνεται. Υπό αυτό το πλαίσιο τέθηκε το θέμα εδώ. Έχουμε πολύ χρόνο λοιπόν να συζητήσουμε και να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα και άλλα θέματα. Σημείωσα σε σχέση με τις ε, προτάσεις ε, για θέματα συμβιβαστικών τροπολογιών που θα πρέπει να εξευρεθούν βάσεις ε, για μια τέτοια προσέγγιση και θα ληφθούν υπόψη αυτά τα θέματα. Ήθελα όμως εδώ για ένα θέμα, ας το πω έτσι, πιστής εφαρμογής αυτών των αρχών να πω τούτο. Έχει δίκιο συνάδελφος τη CCR όταν λέει ότι όταν έχουν αναφερθεί κάποιες τροπολογίες που θα υποβληθούν από την ομάδα του και ότι δεν καλύπτονται λέει από συμβαστικές τροπολογίες κάποια θέματα. Όταν εγώ έθεσα τις τροπολογίες αυτές είδα ότι κάποια θέματα ήταν αντιφατικά σε σχέση με μια συμβαστική τροπολογία ε, ή θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτήν ή όχι. Δεν είναι το ότι το περιεχόμενο το πολιτικό συμπεριλαμβάνεται αυτόματα ή όχι, έχετε δίκιο. Αλλά ήθελα να κάνω αυτή την αναφορά λοιπόν, για να μην μείνει αυτό, ας το πω έτσι, αδιευκρίνιστο για το τι πράγμα κάνουμε λόγο. Αλλά προφανώς σε αυτή την κατεύθυνση ήταν το θέμα αυτό για την αντιφατικότητα. Και για το θέμα του πώς μπορούμε λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε. Όπως και να έχει το πράγμα, οπωσδήποτε είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσω μαζί σας και για τα θέματα διαφάνειας όπως ε, είπαμε. Και για οποιαδήποτε τοποθέτηση θα ήθελα να πω ότι θα είμαι ε, ανοιχτή σε διμερείς τέτοιες επαφές και συναντήσεις και προσβλέπω στο σύντομα να μπορέσουμε να έχουμε μια νέα συνάντηση με όλους τους σκιώδεις εισηγητές για να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο σε αυτή τη διαδικασία. Και ευχαριστώ αν θα μπορούσατε να αποστείλετε τα σχόλιά σας ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το δυνατόν πιο γοργά. Και πάλι για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ματίας. Πάμε στο επόμενο θέμα τη σημερινή σα διάταξη, στο σημείο 8, παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεω για τα ούσιτς. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Σβέν Γκίκολτ. Έχετε το λόγο. So, Θερμά λοιπόν, καλώ ήρθατε. Και είναι ωραίο, μια και πάει κάποιος χρόνος από τότε που το δρομολογήθηκε αυτή η έκθεση, ότι τώρα μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Την πρότασή μου την κατέθεσα ήδη και αδειμονώ να δω ποιε θα είναι οι αντιδράσει των συναδέλφων σε αυτή την έκθεση. Θέλω να επικεντρωθώ σε κάποια σημεία, αν γίνεται. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμπεριέχει καταρχήν τρία θεματικά πλέγματα κυρίως. Πρώτον το θέμα της ευθύνης, της υπευθυνότητας. Δεύτερον το θέμα των κυρώσεων ή προστήμων. Τρίτον τον τομέα των αμοιβών ή αντισταθμιστικών αμοιβών. Είναι σαφές ότι υπάρχει και ένα άλλο πλαίσιο εδώ, το οποίο εντάσσεται στην χρήση usage funds, που αφορούν τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα εμπλέκονται με την απελευθέρωση, φιλελευθεροποίηση αυτού του τομέα τα τελευταία, το τελευταίο διάστημα. Έχουμε και την κατάσταση το ότι εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα έκτο τέτοιο ε, πλαίσιο σε σχέση με το πέμπτο και Μπορούμε όμως ε, να περιοριστούμε και να δούμε, να έχουμε μια συντομότερη έκθεση, εν πάση περιπτώσει, πιο περιεκτική, Όσον αφορά τον τομέα της ευθύνη ε, ή της υπευθυνότητα, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια καλή πρόταση που τους καταναλωτές τους προστατεύει από κινδύνους που προηγούμενα δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν ή να ανοιχνευτούν όπως όταν έχουν κάποιες τέτοιες διαχειριστικές εταιρείες κάποια προβλήματα τότε στο μέλλον διαφορετικά θα γίνεται ή θα αντιμετωπίζεται το θέμα. Οι καταναλωτές θα προστατεύονται σε αντίθεση με το παρελθόν. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυτές οι διατάξεις και αυτοί οι κανονισμοί σε κάποιες ειδικέ περιπτώσεις, σε κάποιες τρίτες αγορές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σε κάποια προβλήματα όταν υπάρχει υποχρέωση για κάποια περιουσιακά στοιχεία ε, ε, να υπάρχει κάποια επένδυση και να χρησιμοποιείται μια τέτοια υπηρεσία και να λένε διαχειριστές τέτοιων κεφαλαίων ότι δύσκολα μπορούν να αξιολογήσουν ποιοι κίνδυνοι ε, συνδέονται με μια τέτοια δράση και πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει να αποκλείονται κάποιες τρίτες αγορές από αυτό το πλαίσιο. Εδώ πιστεύω ότι ως συνάδελφοι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, να δούμε μια λύση ασφαλιστική, ασφαλή, ασφάλειας θα μπορούσε να λειτουργήσει, ασφαλιστικού περιεχομένου. Θυμάμαι ότι η συνάδελφος Περβάος Μπερές είχε προτείνει κάτι τέτοιο σχετικό. Όταν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι, συγκεκριμένοι ε, κίνδυνοι που μέσα από ένα αυστηρό καθεστώς για τη ρύθμιση της ευθύνης ε, δημιουργούν κάποιες επιπτώσεις ανεπιθύμητες, και επειδή πραγματικά δεν είναι αποδεκτό κάποιους από αυτού, τους κινδύνους αυτούς όπως κάποιοι από τους, τις, τους βιομηχανικούς επιχειρησιακούς κύκλους προτείνουν να τους μεταθέσουμε τους κινδύνους στους καταναλωτές τότε αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν υπό τη σύναψη μιας ασφαλιστικής σύμβασης μέσω μιας ασφαλιστικής εταιρείας ώστε να μην επομίζεται κινδύνους που δεν μπορεί να αξιολογήσει ο επενδυτής και από την άλλη πλευρά όμως να υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο θα εντάσει σε αυτό τους κινδύνους αυτούς σε σχέση με ε, κάποιες αγορές. Το δεύτερο θέμα όσον αφορά τα πρόστιμα ή κυρώσεις, ε, την ίδια συζήτηση το, την είχαμε και για την κατάχρηση θέσης στην αγορά ε, που είχε διαξαρθεί και για την οδηγία για τα ίδια κεφάλαια. Προτείνει εδώ και σωστά νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέτοιου είδους κυρώσεις και διοικητικού χαρακτήρα αλλά και ποινικού χαρακτήρα και ποινικέ τέτοιες κυρώσεις ή πρόστιμα πρέπει να εναρμονίζονται και έτσι όσον αφορά κινητά αγαθά όπως assets να μπορούν να ε, λειτουργήσουν. Βλέπουμε ότι στο Συμβούλιο αντιμετωπίζει αντίσταση αυτή η πρόταση, αλλά δεν βλέπω κανένα λόγο να παρεκκλίνουμε από τον προσανατολισμό, από τις κατευθύνσεις που ακολουθούμε για την έννοια εσωτερική αγορά. Το τρίτο που αφορά και τις δικές μου προτάσεις αφορά την ε, αμοιβή τι γίνεται εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχει σχετικά απλά διαμορφώσει τα πράγματα. Ουσιαστικά τους κανόνες που για το IFM είχαμε προβλέψει, δηλαδή τύπου IFM που ουσιαστικά από πλευράς αγοράς ένα στενότερο κύκλο πελατών, σε ένα στενότερο κύκλο, μικρότερο κύκλο στοχεύουν, έχει αντιγράψει πολλά πράγματα και οι περισσότερες ε, διατυπώσεις είναι κυριολεκτικά ένα προς ένα αντιγραφή αυτών των διατάξεων σε σχέση με το ε, Συμβούλιο ε, Κινδύνου, Συστημικού Κινδύνου. Όμως υπάρχουν και κάποια προβλήματα μεταφοράς ή μετάθεσης που έχουν παρισφρήσει εδώ. Και αυτό που κάνω εγώ στην έκθεσή μου είναι προτείνω τους κανόνες του FSB για το θέμα της ε, αποζημίωσης ή αμοιβή να τους μεταθέσουμε, να τους μεταφέρουμε πλήρως, 100%. Και εδώ να δούμε και το θέμα του επόπτη που θα επομίζεται την εφαρμογή αυτών των κανόνων ε, κατά σε σχέση όμως με κάτι που παρατήρησα είναι ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα δεν θα είναι τα θέματα αμοιβή των ίδιων των αρμόδιων, αλλά της αμοιβή των εταιριών αυτών συνολικά, όχι ατόμων. Ακούσαμε από, σε σχέση με ενώσεις προστασίας καταναλωτών, αλλά και από άλλους εμπλεκόμενους το ότι ο τρόπος αμοιβή το της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων πολλές φορές είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί. Έχουμε ταμεία που χάνουν αξία όσο αυτά τα κεφάλαια που διαχειρίζονται, όμως παίρνουν πριμ και, και παίρνουν, ε, ε, ανταμείβονται κιόλας και έχουμε και ταμεία που χάνουν τα κεφάλαιά τους και όμως αξιολογούνται αν έχουν κάποιο όριο το οποίο κάλυψαν ή όχι ως benchmark, ως ορόσημο, ως ε, στοιχείο το οποίο καλύφθηκε. Να πάρουμε ένα γενικό αφηρημένο παράδειγμα για να μην ε, υπάρξει κάποια συγκεκριμένη αναφορά σε επιχειρήσεις. Ένα παράδειγμα, ένα ταμείο επενδύει για παράδειγμα σε equities και παίρνει ως benchmark το MSCI World. Και μετά όμως ταυτόχρονα υπάρχει ένα μίξ, ένα μείγμα αναδυόμενων χωρών που χρησιμοποιούνται, που επενδύονται στα, στις δικές τους μετοχές ή στα δικά τους ομόλογα χρήματα. Είναι τόσο ε, μικρές αυτές οι υποσημειώσεις ε, ως στοιχεία που αθέμητα μπορούν να δίνουν και τη δυνατότητα να αμείβονται για τη διαχείρισή τους αυτά τα ταμεία έχουν ήδη κίνητρο αυτοί να εργάζονται με αυτόν τον τρόπο. Έχουν ροές κεφαλαιακές και μέσω των κεφαλαιακών ροών αυξάνεται και η αμοιβή των ε, υπεύθυνων για τη διαχείριση αυτών των κεφαλαίων, αυτών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τώρα, το να υπάρξουν και κάποια πρόσθετα στοιχεία ως benchmarks τα οποία θα εντάσσονται είναι αμφισβητήσιμη υπόθεση. Για την προστασία των καταναλωτών δεν νομιμοποιείται κάτι τέτοιο, είναι αθέμητο. Γι' αυτό προτείνω στην έκθεσή μου εγώ αυτού του είδους ε, να, ε, πρακτικές να, εκπνε, να λήξουν, να, να μην ε, χρησιμοποιούνται. Και αν θέλουν να κερδίζουν περισσότερα, ε, τότε θα πρέπει να προσελκύουν περισσότερα κεφάλαια τέτοιου είδους εταιρείες. Είναι όμως πολύ δύσκολο να έχουμε με την σωστή διαμόρφωση benchmarks τη διαμόρφωση των αναγκαίων κινήτρων. Πρέπει να υπάρξει η εμπιστοσύνη σε σχέση με τους επενδυτές από τη δράση τέτοιων εταιριών. Αυτό θα ήταν εκείνο το οποίο θα αποκαθιστούσε την εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδου ε, συναλλαγέ. Είμαι βέβαιο ότι με αυτή τη συζήτηση, αυτή τη συζήτηση θα τη συνεχίσουμε, θα τη διεξαγάγουμε με του σκιώδει εισηγητέ. Και αδειμονώ να δω τι γίνεται σε σχέση με εκθέσει σε, σχέση με άλλε αγορέ για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, όπου ω ήθιστε οι περισσότεροι χρήστε ε, έχουν συγκεκριμένη ε, ας το πω τοποθέτηση και συμπεριφορά σε σχέση με τις επενδύσεις τους και δεν δίνουν ε, ουσιαστικά ε, δεν εμπιστεύονται τέτοια κεφάλαια στα χέρια τέτοιων επενδυτών. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι προσβλέπω στη συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές. Να σας αναφέρω και κάτι άλλο ακόμα τώρα ότι ευθύ εξ αρχής είχαμε την πρόθεση να δημιουργήσουμε μια, έναν τομέα εδώ που θα έχει μια συγκεκριμένη ε, οικολογική ας το πω τάση ε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν έχω υποβάλει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, διότι για τα κοινωνικά περιβαλλοντικά θέματα θα εξεταστούν αυτά, αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από πλευρά τη έκθεση περβάσου Μπερέστα θα υπάρχει ευκαιρία να δούμε αυτά τα θέματα. Δεν υπήρχε προτεραιότητα μέσα στο πλαίσιο αυτό το Usage 5 να ενταχθούν αυτά τα κοινωνικο-περιβαλλοντικά θέματα. Δημορώ να ακούσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Muchas Ευχαριστώ κύριε Γκέμπιο. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο συντονιστής ο κύριος Γκοζές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω αρχίσει να λειτουργώ υπερβατικά, μιας και οι συνάδελφοί μου ε, ασχολούνται με άλλες ε, συνεδριάσεις, μου αφήνουν πάντα τα χαρτιά τους για να τα διαβάσω. Λοιπόν, Καταρχά θέλω να ευχαριστήσω τον Σβέν για την προσπάθεια την οποία έχει κάνει. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι τα usage και το FMD έρχονται εδώ να αλλάξουν μια κατάσταση η οποία σε ορισμένους φαινόταν κάπως ε, <clears throat> περίεργη. Οι ρυθμίσεις της οδηγία για τους διαχειριστές των εναλλακτικών ταμείων ε, μερικές φορές δημιουργούσαν προβλήματα σε σχέση με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της usage 4. Ε, το usage 4 είχε γίνει δεκτό πριν γνωρίζουμε τις κομπίνες του Μάντοφ, ενώ η οδηγία που ακολούθησε φυσικά έγινε μετά ε, την περίπτωση του Μάντοφ και αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο τελικά για να υπάρξει μια κάποια προστασία των επενδυτών. Είναι αλήθεια ότι αυτά τα usage λοιπόν είναι ουσιαστικά προϊόν α, λιανικών προϊόντων, προϊόντων λιανικής. Και είναι κάτι το οποίο στην ουσία θέλει να δώσει εμπιστοσύνη εκ νέου στους, στους επενδυτές τους μεμονωμένους. Αν και από ό,τι φαίνεται τα usage δεν, οπεκά αν θέλετε, δεν έχουν υποφέρει και πάρα πολύ από την κρίση και νομίζω ότι αυτή η ετικέτα, η ετικέτα usage, η ευρωπαϊκή ετικέτα κάνει καλό γενικά. Δεν θα πρέπει όμως να είμαστε υπερβολικοί. Στα πλαίσια της συζήτησης η οποία θα ακολουθήσει και στα πλαίσια των προτάσεων των ΜΕΝ και των ΔΕ θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια πραγματιστική και λογική λύση. Δεν θα πρέπει να παίρνουμε σαν παραδείγματα κάποιες ακραίες περιπτώσεις που υπάρχουν σε όλους τους τομείς για να θεωρήσουμε ότι όλος ο τομέας έτσι λειτουργεί και ότι θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις επί τη βάση αυτών των ακραίων περιπτώσεων. Δεν αναφερόμαστε σε ποινικέ διαδικασίες οι οποίες έχουν σαν στόχο να υποστούν κυρώσεις αυτοί οι οποίοι αποκλίνουν παρανόμως. Όχι, να ρυθμίσουμε κάποιες χρηματοοικονομικές συναλλαγές οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από τη βέλτιστη δυνατή ισορροπία ανάμεσα στην απόδοσή τους από τη μία, στην δυνατότητα προσέλκυσης επένδυσης από την άλλη και ταυτόχρονα να δώσουμε στους επενδυτές μια πραγματική αίσθηση ασφαλείας, κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε να έχουμε στο παρελθόν και να μην συμβούν πράγματα τα οποία είχαμε ζήσει παλαιότερα. Γι' αυτό λοιπόν έχω κάθε εμπιστοσύνη στον Σβέν να καταλήξει στη σωστή ισορροπία. Οι εμπειρίες τις οποίες έχουμε από αυτόν δείχνουν ότι είναι ικανός προς την κατεύθυνση αυτή έτσι ώστε και η πρόταση της Επιτροπής που είναι ήδη ικανοποιητική να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω. Ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών δεν ξέρω ποιος θα λάβει τον λόγο. Κύριε Σάιμον παρακαλώ. thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε μιλώντας εκ μέρους της Ελίν Μακάρθη που δυστυχώς είναι άρρωστη και δεν μπορεί να έρθει. Θα σας δώσω πληροφορίες σχετικά με το ποιες είναι οι απόψεις της για το κείμενο. Θέλει να ευχαριστήσει καταρχάς τον εισηγητή, τον κύριο Γκίγκολτ, για την έκθεσή του και αν γέννη καλωσορίζει τις αλλαγές που έχει επιφέρει στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτερα υποστηρίζει τις αλλαγές εκείνες που αφορούν την αμοιβή των managers και τις διατάξεις για την ενίσχυση του καθεστώτος κυρώσεων σύμφωνα με το κείμενο της Επιτροπής για τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς. Υποστηρίζει και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή για να συμπεριλαμβάνονται όλοι εκείνοι που λαμβάνουν αποφάσεις στο, στα usage. Το ευρωπαϊκό μοντέλο usage κατά την άποψή της αποτελεί επιτυχία και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συνέχεια αυτού και την αξιοπιστία αυτού υπό το φως της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσεως Κατά την άποψή της είναι σημαντικό οι επενδυτές να έχουν ασφαλείς διόδους επενδύσεων μέσω των ταμείων usage. Στην παρούσα κρίση θα πρέπει να είναι ασφαλείς οι επενδύσεις στην ευρωπαϊκή πραγματική οικονομία και πρέπει να ενθερρυνθεί, ε, οι επενδύσεις και ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων. Για να συνεχιστεί η εξοπιστία των usage, οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτοί που παίρνουν τι αποφάσει όσον αφορά τις επενδύσεις τους είναι αξιόπιστοι είναι, μπορεί να υποστούν κυρώσει αν ακολουθεί στρατηγικέ παρακινδυνευμένε. Η διαφάνεια και ο έλεγχο και οι αποκαλύψει είναι κάτι βασικό για να γνωρίζουν οι επενδυτές ενδεχόμενου κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Το πακέτο usage θα πρέπει, τα usage πρέπει να δίνουν πλήρε πληροφορίες στους επενδυτές και θα πρέπει να αποκαλύπτονται ε, επίσης και ποια είναι τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν στη διάθεσή τους. Τις επόμενες εβδομάδες θα συζητήσει με τους Σκιώδης ε, τα διάφορα θέματα, τις διάφορες τροπολογίες και προσβλέπει σε αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάιμον. Τώρα για τους φιλελεύθερους, για τον εισηγητή, για την κυρία Χέντσεν, ο κύριος Δίκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι σήμερα μια αξιοπρόσεκτη συνεδρίαση, λέει ο κύριος Κλίντς, γιατί όλο εκπρόσωποι των σκιωδών εισηγητών παίρνουν λόγο. Αυτό δεν συσχετίζεται με το ότι δεν υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον για αυτό το θέμα, που είναι πράγματι πολύ σημαντικό, διότι τα θέματα αυτά από τότε που ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα έχουν μεγάλη σημασία για τα ΟΣΕΚΑ και θα πρέπει να τηρηθεί αυτή η κατεύθυνση και να γίνει το αναγκαίο ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και να αποτραπούν οι κίνδυνοι από τέτοια προϊόντα. Ο Ζαν Πολ Γκοζές ανέφερε την περίπτωση Μέντοφ, που αφορά ιδιαίτερα και τα, τα θέματα το, της χρήσης αυτών των κεφαλαίων. Χρησιμοποιήσαμε αυτή τη δυνατότητα με το Usage 4. Αν θα είχαμε ένα τέτοιο διαβατήριο, ένα τέτοιο πιστοποιητικό για αυτά, ένα κύριο θέμα σε αυτά τα θέματα είναι ε, η ευθύνη αυτών των ε, ιδρυμάτων ή τραπεζών και το ανέφερε και ο Ζαμπόλ και είναι πρόδειλο να πει κανείς ότι το καθεστώς ευθύνης μπορεί να προσανατολίζεται σε σχέση με εκείνο που έχουμε για το IFM. Παρότι πρέπει να ομολογήσω ότι εδώ ουσιαστικά έχουμε ένα προϊόν μπροστά μας που τους μικρούς ε, επενδυτές αφορά περισσότερο σε σχέση με τους μεγάλους. παρόλα αυτά θα πρέπει να ε, στοχεύσουμε στην κατεύθυνση που ανέφερα πιο πριν. Αυτό θα ήταν σκόπιμο. Τώρα, η διεύρυνση των επιλέξιμων ε, ταμείων από πλευράς των ε, ταμείων διαχείρισης και το κατά πόσον αυτό εμπλέκεται στις merger markets, σε συγχωνεύσεις ή σε τέτοιου είδους συναλλαγές, ο επενδυτής θα, μπορεί, θα πρέπει να γνωρίζει σαφώς αυτή την πτυχή. Εγώ εκπροσωπώ την κυρία Άννα από την ε, Δανία. Κάποιες σημειώσεις μου άφησε και τις έχω εδώ που επιλέξει θα σας διαβάσω κυριολεκτικά στα αγγλικά τα παραθέματα σε τρία ε, τμήματα. Sanctions και Remunerations. Έχουμε λοιπόν σαν, γενικό, γενική αρχή ότι δεν μπορεί να είναι διαχειριστής σε μια τράπεζα και ταυτόχρονα να είναι ε, αποθέτης. Θα πρέπει να υπάρξει διαχωριστική γραμμή εδώ. Αυτό το οποίο δεν αντιμετωπίζεται είναι σε σχέση και με τα αποθετικά κεφάλαια αυτά δεν υπάρχουν σαφείς ε, κανονισμοί ποιου είδους ε, ε, ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Στη σημερινή οδηγία είναι ασαφές σε ποια καθήκοντα θα έχει ένας αποθέτης όταν θα πρέπει να επιλέξει νομισματικά ένα τέτοιο είδος επένδυσης. Δημιουργείται μια νομική αβεβαιότητα σε σχέση και με πιθανές απώλειες, απώλειας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα οικονομικά ιδρύματα ε, μπορούν να έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Οι ε, συμβολεογράφοι μπορούν μόνο ως ε, διαμεσολαβητές να δράσουν. Μετά από τα όσα έγιναν το 2001 και σε σχέση με τη διεύρυνση των αποθεματικών αυτών, η ανάγκη αυτή για την ρύθμιση καθίσταται σαφής θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορεί να επιλέγει κανείς ένα τέτοιο διαμεσολαβητή σε τρίτη χώρα. Εδώ ακολουθείται από κάποιους ένα αυστηρό ε, καθεστώς, αν υπάρξουν απώλειες, τότε ο αποθέτης ε, πρέπει να καλύψει τις απώλειες αυτές. Έχουμε λοιπόν διαφορές ε, που δημιουργούνται σε σχέση με κράτη-μέλη μεταξύ τους. Η ανακοίνωση της 9 η Δεκεμβρίου 2010 ενισχύοντας το καθεστώς κυρώσεων στον οικονομικό τομέα μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί σε διάφορες ε, εκθέσεις ε, π.χ. για την οδηγία ε, καταχρηστικού ρόλου στις αγορές και αυτό καθιστά αναγκαίο να, επαν, να προσαρμοστούν τα εθνικά καθεστώτα όσον αφορά το καθεστώς κυρώσεων. Οι διαφορές σε οικονομικού είδους, ε, ε, ε, στο βαθμό κυρώσεων, με διαφορετικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται σήμερα για τις διοικητικές τέτοιες κυρώσεις και τις διαφορές που δημιουργούνται, ο Σβεν Γκίγκολτ ανάλωσε πολύ μεγάλο χρόνο από το έργο που επετέλεσε για το θέμα των αμοιβών των διαχειριστών και πολλές φορές ε, με βάση τα κέρδη αμείβονται αυτοί. Αυτή η κατάσταση κάνει πολλούς από τους διαχειριστές πολλές φορές να υπομίζονται υπερβολικούς κινδύνους ε, στις επενδυτικές δραστηριότητες τους. Είναι λοιπόν δικαιολογείται ότι πρέπει να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές ε, που συστήνουμε να ακολουθηθούν. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κύριε Κλίντς. Εξ ονόματος φέρω κύριος Καμάλ παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω την έκθεση του ΣΒΕΝ. Ε, αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, λοιπόν, δεν ξέρω ποια μεγαλύτερη πρόκληση από τα θέματα που έχουν συζητήσει. Θα είναι επιτυχής, πιστεύω, σε όσε προσπάθειε που καταβάλει ο ΣΒΕΝ. Είναι καλό που βλέπουμε ότι υπάρχει αναφορά σε άλλους κανονισμού και οδηγίε. Εδώ θέλουμε να επικαιροποιήσουμε τον κανονισμό και τις άλλες προτάσεις να λαμβάνουμε υπόψη. Όσον αφορά την ευθύνη του αποθέτου, ε, έχω κάποιες ανησυχίες. Συμποστηρίζω την άποψη ότι πρέπει να είναι σαφές ε, ποιο, πού σταματάνε οι ευθύνε. Είναι ενδιαφέρον. Ε, όλοι ανέφεραν το φάσμα του Μάντοφ πάντα στις συζητήσεις. Ποτέ δεν είπε ότι ήταν hedge fund όμως. Λοιπόν, και χαίρομαι που σωστά τίθεται διάφορα θέματα στην έκθεση. Λοιπόν, αν υπάρχει παράξενη δραστηριότητα, υπάρχει συνένεση, δεν υπάρχει διαφορά στον αφορά ότι κάποιο είναι υπεύθυνο. Και έτσι πρέπει να είναι. Γι' αυτό το usage 5 πρέπει να προσαρμοστεί με άλλε ρυθμίσει σχετικέ. Το θέμα είναι αν θέλει ο αποθέτης να απαλλαγεί νομικά των ευθυνών του. Χαίρομαι που ακολουθεί ανοιχτή προσέγγιση όσον αφορά τι επενδύσει των αναπτυσσομένων χωρών. Διότι ο ομόλογο σου ε, ε, ε, πρέπει να είναι σίγουρος Κάποτε μου λέγανε ότι δεν, ήθε, δεν θέλαν σε πρώτερε συζητήσει να αναφέρονται αναπτυσσόμενε χώρε και γι' αυτό χαίρομαι που είσαι ανοιχτή προσέγγιση όσον αφορά. Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι το εξή. Ένα διαχειριστή ταμείου, ένα ε, πελάτη θέλει να επενδύσει στην απτυσσόμενη χώρα. Αλλά ο αποθέτη ε, έχει ανησυχίες. Δεν θέλει να λάβει τον κίνδυνο το ταμείο. Δεν θέλει την ευθύνη. Το θέμα είναι ότι αν διαχειριστή του πόρου επιμένει στην επένδυση, τότε φέρει πάντα ευθύνη ε, ο αποθέτη. Θα πρέπει να βρούμε τη λύση να μπορεί ο αποθέτης αυτές τις περιπτώσεις να απαλλαγεί τον ευθυνών του, να επιτρέψει στον επενδυτή να επενδύσει σε αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά να υπάρχει ευθύνη κάποιου. Κάποιος πρέπει να υπομειστεί την ευθύνη στο τέλος. Είναι δίκιο να περιμένουμε αποθέτης να έχει την ευθύνη όταν εκείνος θα είχε αποθαρρύνει την επένδυση. Και αν έχουν την ευθύνη, μπορεί να σταματήσουν και τι επενδύσει στι αναπτυσσόμενε χώρε. Πρέπει να ενθαρρύνουμε όμω τέτοιε επενδύσει στι αναπτυσσόμενε χώρε στο μέτρο του δυνατού. Όσον αφορά τι αμοιβέ, έχω κάποιε ανησυχίε. Όταν είχαμε συζητήσει στο CRD3, θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει οι τραπεζίτε και οι διαχειριστέ αυτών των πόρων να έχουν τη διαμοιβή. Διότι δεν αντιπροσωπεύεται ο ίδιο συστημικό κίνδυνο. Είναι διαφορετικά τα επιχειρηματικά μοντέλα. Πιστεύω ότι θα πρέπει η αμοιβή να αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις. Δεν χρειάζεται ανώτατα όρια όσον αφορά τα μπόνους. Χρειάζεται εξορθολογική προσέγγιση. Έχουμε συζητήσει και σε άλλες περιπτώσεις τις αμοιβέ. Και έχουμε κάνει και ακολουθήσει και τον Ιανουάριο έχουμε δημοσιεύσει κάποιες κατευθύνες γραμμές. Οπότε η συζήτηση πρέπει να είναι λογική, να ευθυγνωστή η προσέγγιση για το usage ε, οι επενδυτές με την αμοιβή εκείνων που χειρίζονται τα ταμεία. Το ECR θα ήθελε να υπάρξει σχετισμός επιδόσεων με αμοιβή. Το θέμα είναι πώς το πετυχαίνουμε. Ήταν πάντα δυνατόν να υπάρξει ευθυγράμμιση της απόδοσης με τις επιδόσεις, αμοιβής με επιδόσεις. Ε, υπάρχει βαθμολόγηση. Πώς θα γίνεται η βαθμολόγηση. Καμιά φορά οι managers πληρώνονται ακόμα και όταν έχουν κακές επιδόσεις. Μπορούμε να πετύχουμε αυτό το σχετισμό. Πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Δεν έχω προκαταλήψεις. Και χαίρομαι που θα συζητήσουμε μαζί, με σένα, που εξετάζει τις συνέπειες των συζητουμένων. Ας το εξηχνιάσουμε. Μπορούμε να συναρτήσουμε αμοιβή με επίδοση ή μπορούμε να καλύψουμε το θέμα διαφορετικά. Πρέπει να προστατεύονται περισσότερο οι επενδυτές. Χωρίς πολλές απαιτήσει και όρους που να έχουν αρνητικές συνέπειες. Προσβλέπω συνεργασία με τον εισηγητή. Ελπίζω να μην μείνει άϊπνος πολλές νύχτες μια και είναι νέος πατέρας αλλά μπορώ να του πω ότι σαν σκιώδης συζητητή δεν θα του δώσω παραπάνω ξενύχτη από ό,τι θα είχε τα παιδιά του. Σας ευχαριστούμε κύριε. Σας ευχαριστούμε. Από την ΚΟΕ δεν υπάρχει κανεί και έτσι ξαναδίνουμε το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Γκίγκολτ. Uh, uh, so first for the... Ευχαριστώ. Καταρχάς, ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα θετικά σχόλια και τα σχόλια γενικότερα. Πρώτον, να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ξέρω αν η μεταφορά των απόψεων του Κανφίν ήταν ε, λίγο σαν καρικατούρα θα έλεγα. Αλλά και οι Γάλλοι υπουργοί είναι υπέρ φυσικά τη συνέχισης των επενδύσεων και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πάντως <clears throat> αυτά τα επενδυτικά σχήματα μπορεί να βοηθήσουν στις επενδύσεις και δεν υπάρχει τίποτα το κακό αν οι επενδυτές θέλουν να παίρνουν μέρος στις αποδόσεις. Πάντως θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση εδώ και εγώ έρχομαι στα σχόλια του Κλίντς. Αν πράγματι θέλει κανείς να διατρέξει ε, κινδύνους έτσι και αλλιώ ε, επενδύοντας σε ε, σχήματα στις αναδυόμενες αγορές. Δεν μπορεί να ελέγξει κανείς αν στο εξωτερικό σε χώρες άλλες ο, αυτός ο οποίος έχει αναλάβει την κατάθεση των τίτλων ε, έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν μπορεί να ελέγξει κανείς ακριβώς το πώς γίνεται στην Βραζιλία και το πώς ε, επενδύονται τα κέρδη από τις αποδόσεις. Αν όμως κάποιος θέλει να διατρέξει τον κίνδυνο να προχωρήσει σε μια τέτοια επένδυση χωρίς να ελέγχει απόλυτα αυτούς τους οποίους έχουν γίνει καταθέσει των τίτλων, γιατί όχι. Ε, το θέμα είναι ο επενδυτής να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους θα αναλάβει, να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους θα έχει να διατρέξει και ανάλογα θα αξιολογήσει την ποιότητα την συγκεκριμένη εταιρεία που έχει αναλάβει ε, την ε, χρήση θα έλεγα των συγκεκριμένων ποσών. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί επί τη βάση συγκεκριμένων ρυθμίσεων για την απόδοση ευθύνης. Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτό είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και μπορεί να οδηγήσει σε αποεμπενδυτικές προσπάθειες, δεν ξέρω ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αλλάζει συνεχώς, ε, θα έλεγα, θέση τελικά. Αν κάτι τέτοιο είναι δικαιολογημένο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης που απομακρύνει τους κινδύνους για τους ε, επενδυτές, γιατί όχι, Αν αναδούμε πώς. Το ίδιο ισχύει και σχετικά με το καθεστώς των κυρώσεων. Αυτά που άκουσα είναι θετικά. Σχετικά με τις αμοιβέ των στελεχών. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι προφανώς και συμφωνώ στο ότι η επίδοση και η αμοιβή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες. Αλλά νομίζω ότι στον τομέα των ταμείων αυτών η σχέση αυτή έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Τα ταμεία μπορεί να δει κανένα ε, τις επιδόσεις, τους πίνακες τους, αυτά που πηγαίνουν καλά έχουν πάρα πολλές εισρωές και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο να αποδώσουν καλά το θέμα είναι η ανάπτυξη του ταμείου για τα στελέχη των ταμείων, γιατί αν τυχόν αυξάνονται τα διαθέσιμα των ταμείων τους, αυξάνονται φυσικά και ε, οι αμοιβέ τους. Αυτό που δεν θα ήθελα να δω εγώ, είναι να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο, το οποίο θα έχει διαμορφωθεί με εντελώς αδιαφανή τρόπο, Ένα άλλο θέμα βέβαια είναι και η κουλτούρα τη λεγόμενη των πόνους. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο στην περίπτωση του CID αποφασίσαμε να το ε, αλλάξουμε. Ξέρω ότι βέβαια είχε δημιουργήσει κάποια προβλήματα, αλλά νομίζω ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν τώρα πια τα μπόνους τα οποία κάποτε υπήρχαν σε τόσο υψηλά επίπεδα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν τμήματα της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας που καλύπτονται από αυτήν την αντίληψη θα έλεγα ε, για τα βραχυπρόθεσμα κέρδη και υψηλότατες αμοιβέ ακριβώς λόγω αυτού του υψηλού επίπεδου των βραχυπρόθεσμων κερδών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Συμφωνώ με αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει. Εμείς ας προσπαθήσουμε να ευθυγραμμίσουμε τις απόψεις μας γύρω από την λογική αυτή στις προηγούμενες εκθέσεις. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με τον τρόπο αυτό και οι πελάτες των usage ε, ε, αξίζουν μεγαλύτερης προστασίας από ότι αν επενέδυαν σε hedge funds σαν παράδειγμα. Όπου και εκεί βέβαια έχουν υπάρξει κάποιες ε, αλλαγές μετά από προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, με μεγάλη χαρά θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με όλους σας και με τον κύριο Καμάλ. Ευχαριστώ Σβέν. Σε αυτή τη φάση λοιπόν θα σταματήσουμε μέχρι τις 5. Το επόμενο θέμα είναι η κοινή συνάντηση με την Επιτροπή Απασχόλησης με τους Επιτρόπους Άντορ και ε, Ρεν. Α, συγγνώμη. Ξέχασα να σας πω ότι η προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών είναι η 17η Δεκεμβρίου. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει την 21η Ιανουαρίου του 2013 και η ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί πότε θα γίνει. Λοιπόν, όπως σας έλεγα προηγουμένως, το επόμενο θέμα είναι στις 5 ακριβώς. Κοινή συνάντηση με τους επιτρόπους Ρεν και Άντορ για τον οικονομικό διάλογο ε, και την ε, έρευνα για την ετήσια ανάπτυξη. Ε,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

You say this is not yet joint meeting. Okay, everybody. Um, Καλώς, καθίστε παρακαλώ. Δεν έχει ξεκινήσει η κοινή συνεδρίαση γιατί περιμένουμε ακόμα τους επιτρόπους. Αλλά από πλευρά της δικής μας επιτροπής δεν έγιναν οι ανακοινώσεις του Προέδρου μέχρι τώρα, της Προέδρου καλύτερα, και γι' αυτό θα τις κάνω τώρα έτσι ώστε να σας διασκεδάσω λίγο. Καταρχάς ο οικονομικός διάλογος με τον κύριο Γιούνκερ, τον πρόεδρο δηλαδή του Eurogroup, Ξέρετε ότι κανονικά έπρεπε να γίνει σήμερα το απόγευμα. Την Παρασκευή ήδη μας είπε ο κύριος Γιόνκερ ότι δεν θα μπορούσε να είναι ανάμεσά μας και γι' αυτό του πρότεινα κάποιες άλλες πιθανές ημερομηνίες το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο για αυτόν τον σημαντικό οικονομικό διάλογο. Όπως γνωρίζετε, θα ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση με τους επιτρόπους Ρεν και Αντόρ, που θα γινόταν αύριο, θα γίνει σήμερα, ε, γιατί ο κύριος Όλη Ρεν δεν είναι διαθέσιμος αύριο. Εν πάση περιπτώσει προσπαθήσαμε να διορθώσουμε μια κατάσταση που δεν ήταν πολύ καλή. Τώρα για τους συνεχιζόμενους τριμερείς διαλόγους για τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει των πιστοτικών ιδρυμάτων. Είχαμε πολιτικούς ε, τέτοιου είδους ε, διαλόγους τριμερείς ε, την Παρασκευή για τον ορισμό του κεφαλαίου, για τα λεγόμενα benchmarking, για τις εσωτερικές αξιολογήσεις. Μια τεχνική συνάντηση έχει ήδη γίνει την προηγούμενη Τετάρτη για να ενσωματωθούν όλες αυτές οι συμφωνίες στις λεγόμενες συμβιβαστικές τροπολογίες. Ο επόμενος πολιτικός διάλογος τριμερής θα γίνει αύριο μετά από την έκτακτη συνεδρίαση της δικής μας Επιτροπής γύρω στις 11. Για το διπλό πακέτο, το Τούπακ, έγιναν συναντήσεις στο προηγούμενο Στρασβούργο και για τις δύο προτάσεις εκθέσεων υπήρξε μια κάποια πρόοδος και για τα θέματα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και για το μνημόνιο κατανόησης και ε, για τη στάθμιση των ψήφων στα πλαίσια της έκθεσης Γκοζές. Για τις εκκρεμότητες στην έκθεση Φεραίρο υπάρχουν ε, ε, τα θέματα των κατεξουσιοδότησης πράξεων, τα θέματα του κεφαλαίου 3, και επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις συνέπειες της ύφεση στα πλαίσια των διαδικαστιών υπερβολικών ελλημάτων που έχουν ξεκινήσει. Όλα αυτά θα γίνουν αύριο. Για τις οίκους αξιολόγησης, ο τριμερής διάλογος ολοκληρώθηκε ε, στις 20 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Μπαρνιέ Έγινε και άλλη μια συνάντηση χθε ε, για τις εκκρεμότητες όπως τα θέματα αξιολόγησης του δημοσίου χρέους. Και τέλος, η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Οικονομικών στην Λευκοσία. Ο κ. Στόλογιαν εκπροσώπησε την Επιτροπή μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης υπήρξε και ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης που ασχολήθηκε με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Ε, ναι, με τα κοινοβούλια των κρατών μελών φυσικά ασχολούνται με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά αναγνωρίζουν οι εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων τις πρωτοβουλίες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για να γίνει μια συνάντηση κοινοβουλευτική για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Να προσθέσω εδώ ότι είχατε επίσης και την έκθεση, ακούσατε την έκθεση από την αντιπροσωπεία στο Δουβλίνο, αλλά είναι θέματα που θα συζητήσουμε και με την επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία, έτσι ώστε να μπορέσουν να μας κρατήσουν ενήμερους γύρω από τα θέματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα με τους δύο επιτρόπους, θα πρέπει να διακόψουμε για λίγο Okay. we will start you You may have noticed. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα παρατηρήσατε ότι έχουμε παρόντα τον Επίτροπο Ρεν. Ο Επίτροπος Άντορ καθυστέρησε λόγω συνεντεύξεως τύπου. Οπότε κινούμεθα με βάρδιες. Θα αλλάξουμε δεόντως και την ημερήσια διάταξη αναλόγως με τους παρόντες επιτρόπους. Καλωσορίζω τον Επίτροπο Ρεν και τον Επίτροπο Άντορ και τα μέλη της Επιτροπής της Οικονομικής και Ομισματικής και της Επιτροπής Απασχόλησης, διότι πρόκειται περί κοινής ε, Οπότε ας, σας ρωτώ αν εγκρίνετε τη μερίσια διάταξη. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Θα υπάρξουν ερωτήσεις για τον Επίτροπο Ρεν πριν ακούσουμε τον Επίτροπο Άντορ. Ε, αν έτσι χρειαστεί να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον Όλη να μας κάνει την παρουσίασή του για ένα δεκάλεπτο. Ευχαριστώ, Σάρα, Σάρον. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω σε ένα δεκάλεπτο τον κόσμο την ευρωπαϊκή οικονομία. Πρόκληση. Κυρίες και κύριοι, έρχομαι από τη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί στις 8. Μετά από αρκετέ εβδομάδες προετοιμασιών και για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση, μετά από εβδομάδες προετοιμασίες για την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη. Πριν από μισή ή μία ώρα τελειώσαμε τη συνεδρίαση. Άφησα τον πρόεδρο Μπαρόσο να δώσει τη συνέντευξη τύπου. Και ο Λάσλο Άντορ, ο συνάδελφος, θα μείνει και αυτός εκεί για λίγο και θα καταφτάσει όταν θα απελευθερωθεί από τη συνέντευξη τύπου. Υπενθυμίζοντα τα όσα είπε ο Ζακ Ντελόρ. Χρειαζόμαστε δηλαδή και και, αρχιτέκτονες και πυροσβέστες για την ευρωπαϊκή οικονομία και αυτή την εβδομάδα εξεπλήρωσα αυτά που είπε ο Ντελόρ. Δευτέρα, Τρίτη ήμουν πυροσβέστης για την Ελλάδα και το τελευταίο 48ωρο εργάστηκα επί των σχεδίων για μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Άρα ανοικοδόμηση των θεμελίων της Ευρώπης με άλλα λόγια. Χαίρομαι που είμαι εδώ και έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω για την, για την ετήσια αυτή έκθεση την έρευνα για την ανάπτυξη που εθετήθηκε πριν από μία ώρα. Και εκεί ε, αναφερόμαστε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέτουμε τις προτεραιότητες για την αιτήσια πολιτική ανάπτυξης και ξεκινά και το καινούριο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα είναι το τρίτο αυτό που θα ξεκινήσει. Είναι πολύ σημαντικό τμήμα οικονομικού διαλόγου για ανταλλαγή απόψεών μας τώρα. Και λαμβάνει χώρα σε πολύ σημαντικό σταυροδρόμι, σε μια καμπή, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που συζητούν το μελλοντικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Πώς θα μεταρρυθμιστεί το πλαίσιο. Παρουσιάσατε τις απόψεις σας εσείς στην έκθεση Tyson. Συζητήθηκε στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο την ε, περασμένη εβδομάδα έγκαιρη και σημαντική συμβολή του Κοινοβουλίου. Εκτιμάται πολύ. Με τα χαρά είδα ότι συμφωνούμε σε πολλούς τομείς. Επίσης ελπίζω ότι θα δείτε ότι αντικατοπτρίζεται αυτή η συμφωνία και στο προσχέδιο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υθετήθηκε σήμερα, όπως προανέφερα. Πριν στραφώ στην επισκόπηση αυτής της ανάπτυξης, να αναφερθώ σε αυτό το σχέδιο για μια εμβάθυνση της ε, Ευρωπαϊκής Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης, μιας πραγματικής ένωσης, που σχετίζεται άμεσα με το Tupac, το διπλό αυτό πακέτο, και που απασχολεί ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. Εκεί, στο σχέδιό μας, καθορίζουμε οδικό χάρτη. Δράσεις που είναι απαραίτητες, βράχη, μέσο, μάκρο πρόθεσμα, για να επιφέρουμε πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Βραχυπρόθεσμα θέλουμε να εφαρμόσουμε τα συμπεφωνηθέντα και να εθετήσουμε όσα έχουν δρομολογηθεί. Το επόμενο εξάμεινο με 18 μήνο. Θέλουμε να βελτιώσουμε και μέσω ε, δευτερογενούς νομοθεσίας το όλο πλαίσιο. Μεσοπρόθεσμα θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε, να επιφέρουμε μεταρρυθμίσεις που συνεπάγονται αλλαγές της συνθήκης. Μακροπρόθεσμα προβλέπουμε μεταρρυθμίσεις που θα απαιτούν πιο θεμελιώδεις αλλαγές των συνθήκων. Καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων θα έλεγα ότι το σχέδιο εξισορροπεί τις μεγαλύτερες ευθύνες με τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη στην Ευρωζώνη. Προτείνονται και διάφορα βήματα για δημοκρατική νομιμότητα και δυνατότητα σωστού ελέγχου, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα σωστή και παρκή ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από πολλές πλευρές αυτό το σχέδιο συνάδει και με την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πραγματική νομισματική ε, ένωση που εξεφράστηκε από το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα στην έκθεση που εγκρίνατε. Έχουμε οδικό χάρτη με χρονικά πλαίσια και προτείνουμε μέτρα για υποστήριξη της ανάπτυξης, βραχυπρόθεσμα. Θα επιτευθεί αυτό μέσω διευρυμένου συντονισμού οικονομικών πολιτικών μέσω συστηματικών εκ των προτέρων ελέγχων και τη δημιουργία, την ανάπτυξη ανταγων, ε, δημιουργία ενός μέσου ανταγωνιστικότητας και σύγκλησης. Εκφράσαμε και την προθυμία να διαρευνήσουμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε επιχειρηματικό χαρακτήρα σε φυστάμενες διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Για να έχουμε επαρκείς επενδύσεις, ούτως ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη μέσω καταλήρων μέσων. Έχουμε εισάγει μέτρα για να ολοκληρήσουμε πραγματική οικονομική και νοσματική ένωση μεσοπρόθεσμα κινούμενη προς ενίσχυση οικονομικής, οικονομικού και πολιτικού συντονισμού που θα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τη μείωση του δημοσίου χρέους σε σημαντικό βαθμό ξεπερνώντας τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δημιουργώντας το Ταμείο Διάσωσης και την έκδοση ευρωμολόγων. Αυτό θα συμβάλλει σε καλύτερη αγορά, ενωμένη αγορά ε, τίτλων στην Ευρωζώνη και θα οδηγήσει στην οικονομική σταθερότητα. Εν γέννη, αυτό το σχέδιο περιγράφει πραγματικά βήματα προς πραγματική οικονομική και ένωση και συμπίπτει αυτό με τις απόψεις του Κοινοβουλίου που αντικατοπτρίζεται στην έκθεσή σας. Δεν θα γίνει εν μία ανοιχτή αυτό. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές για τα πολιτικά όρια που υπάρχουν. Εστέ βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστεί άοκνα από αυτού και ελπίζω ότι αυτή η δέσμευση που αναλαμβάνουμε θα οδηγήσει σε μια συμφωνία όσον αφορά το, το πακέτο, το διπλό πακέτο, το πακέτο με τα δύο μέτρα που θα θετήσουμε, το 2 Όσον αφορά τις άλλες προτεραιότητες της επισκόπησης αυτής για την ανάπτυξη της έκθεσης, να τονίσω τρεις βασικούς τομείς που εξετάσαμε από τους πέντε. Και ο Λάζλο Άντορ, πιστεύω, θα ασχοληθεί με την απασχόληση και την αντιμετώπιση της μεγάλης ανεργίας. Συνεργαζόμαστε στενά για αυτά τα ζητήματα με τον Λάζλο. Καταρχάς, πρέπει να ολοκληρώσουμε ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση του χρηματοστητικού τομέα. Δεν πρόκειται περί διασώσεως τραπεζιτών. Πρόκειται περί εξασφαλίσεως τη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που συνιστούν την πραγματική οικονομία, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βελτιωμένη η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις εταιρείε μας είναι ουσιαστικό, ουσιώδες για την ενίσχυση της εξαγωγής και της βιομηχανικής παραγωγής. Πρέπει να ενισχύσουμε την επένδυση του δημόσιου και του ιδιωτικού ταμέα για να κινηθούν οι τροχοί της ευρωπαϊκής οικονομίας εκ νέου. Γι' αυτό η αύξηση του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του κεφαλαίου διάσωσης που αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατόπιν πρότασής μας, θα είναι κάτι που ήδη θα αντικατοπτρίζεται στο δανειοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Ανάπτυξης από τον επόμενο χρόνο 180 δισεκατομμύρια ευρώ θα ιδρυθούν για επενδύσεις την επόμενη τριετία για καινοτομία και δεξιότητες, πρόσβασης μικρομεσών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, στρατηγικές υποδομές και αποδοτική χρήση των πόρων. Μετά θα πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας προς διαθετικές αλλαγές, διαθετικές μεταρρυθμίσεις και σχετικά με αυτό έχουμε δρομολογήσει κύμα μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Ισπανία, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλον, να διευκολυθούν οι επιχειρηματίες, να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις και να μεγαλώσουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις. Πρέπει να δούμε και τις επιδόσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και ποιες και να υπάρχουν και καλύτερες δεξιότητες. Πρέπει να επενδύσουμε στους εγκεφάλους της Ευρώπης για να ανταγωνιστούμε παγκοσμίως και φραγμή για τον ανταγωνισμό στον τομέα της ενέργειας και του ανταγωνισμού είναι κάτι που θα πρέπει να καταπολεμηθεί, να διερευνηθεί. Πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα των δημοσιονομικών με εξυγίανση των οικονομικών που θα πραγματοποιηθεί με ευφύ τρόπο. Άρα θα πρέπει να διατηρηθούν οι επενδύσεις σε τομείς που είναι απαραίτητοι για τη μελλοντική ανάπτυξη, όπως έρευνα, καινοτομία, παιδεία, ενέργεια. η ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση εξακολουθεί να δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο ούτως ώστε τα δημοσιονομικά να επανέλθουν σε βιώσιμα επίπεδα και να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις που ισχύουν σε κάθε χώρα. Όπως προανέφερα, είναι σημαντικό το σύμφωνο, θα θέλαμε να πούμε το σύμφωνο σταθερότητας ανάπτυξης δεν είναι κάτι ανόητο, αλλά εστιάζεται επί των ελλείψεων των υποδομών. Πρέπει να εξετάσουμε πώς κινείται και ο οικονομικός κύκλος. Γι' αυτό εστιαζόμαστε επί των διαφορετικών οικονομικών προσπαθειών που γίνονται από κάθε χώρα όταν εξετάζουμε τη συμμόρφωσή τους, όχι μόνο επί ονομαστικών ε, στόχων, παρόλο που είναι πηχαίοι τίτλοι στα μέσα ενημέρωσης αυτή η στόχη. Δεν εστιαζόμαστε όμως μόνο σε αυτό να σας πω ότι ήδη στο σχέδιο είναι, αλλά είναι κάτι που έχει άμεση σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και την εξυγίανση. Θα διερευνήσουμε και άλλους τρόπους εντός των ισιών των κανόνων και το συμφώνου, ούτω ώστε να συμπεριλάβουμε και τα πενδυτικά προγράμματα στην αξιολόγηση των προγραμμάτων ε, σύγκλησης και ανάπτυξης. τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων που βελτιώνουν τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών. Θα μπορούν να εξαιρεθούν προσωρινά από τους μεσοπρόθεσμους στόχους. Κρατικές επενδύσεις και προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη. Κάτι που ταιριάζει με την αντιξιακή μας πολιτική και με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι, για να κλείσω, θα ήθελα να πω ότι προχωρήσαμε πολύ τα τελευταία δύο-τρία χρόνια προσπαθώντας να μεταρρυθμίσουμε την οικονομική διακυβέρνηση. Πρέπει να ξεκολουθήσουμε να προσπαθούμε για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Και αυτές οι αιτήσει εκθέσεις ανοίγουν το δρόμο για τέτοιες πολιτικές που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να επανέλθει στην ανάκαμψη του χρόνου, να ενισχυθεί η ανάκαμψη και η οικονομική ε, ανάπτυξη την επόμενη περίοδο, ούτως θα διευκολύνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την συνεχιζόμενη οικονομική εξυγίανση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μας λείπει πάντα ο κύριος Σαντόρ, μιας και αυτός ε, σας αναπληρεί ουσιαστικά στη συνέντευξη τύπου, θα τον αναπληρώσετε κι εσείς εδώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στους εισηγητές της κάθε επιτροπής για την ε, έρευνα για την ετήσια ανάπτυξη. Πρώτα, η κυρία Φεραίρο από την Επιτροπή ΕΚΟΝ και μετά η Βερόνικα από την Επιτροπή Απασχόλησης. Θα μιλήσω την Αγγλική, λέει και κυρία Φεραίρα. Προετοιμάζουμε τη νέα έκθεση. Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε ότι το Κοινοβούλιο έχει ένα επιπλέον ρόλο να παίξει στα πλαίσια αυτής της συζήτησης. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε την κρίση μέχρι τώρα. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, επαναλαμβάνω. Η στρατηγική σταθεροποίηση απέτυχε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια τεράστια προσπάθεια να ανοιχνεύσει κάποια ίχνη ανάκαμψης στις χώρες οι οποίες πειθαρχικά ακολουθούν τις συστάσεις της. Στην ουσία όμως και με πραγματικούς αριθμούς οι προσπάθειες λιτότητας ακολουθήθηκαν από κάποιες χώρες υπάκουες και από κάποιες λιγότερο υπάκουες. Οι προσπάθειες λιπρότητας έφτασαν σε υψηλότατα επίπεδα. Έχασε η Ελλάδα 18 πόντους στα έπ 6,5 στην Ισπανία, 4,5 στην Ιταλία και τα αποτελέσματα που είναι. Η λιτότητα οδηγεί σε μια ολοένα αυξανόμενη ύφεση οι προβλέψεις συνεχώς αναπρογραμματίζονται προς τα κάτω βέβαια. Οι συνταγές μέχρι τώρα στην ουσία μας οδηγούν σε μια συνεχή διαδικασία ύφεσης. Οι προοπτικές για το σύνολο της Ευρωζώνης είναι αρνητικές για τον επόμενο χρόνο και θα είναι αρνητικές και για φέτος βέβαια. Τα spreads φυσικά συνεχίζουν να αποκλίνουν η ανεργία έχει φτάσει σε εκρηκτικά επίπεδα. Η μισή από τους νέους σε αρκετές χώρες δεν έχουν μέλλον πλέον στον τομέα της απασχόλησης. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Οι πολίτες δεν μπορούν να επιβιώσουν με μια στρατηγική η οποία δεν αποδίδει. Οι λαοί δέχονται τις θυσίες εφόσον θεωρούν ότι κάπου θα τους οδηγήσουν θα πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, θα πρέπει και εσείς να αποδείξετε ότι έχετε δίκιο, θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί. Έγινε μια μελέτη από τρία πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το UFCE από τη Γαλλία, με το Δανέζικο και το IMK από τη Γερμανία παρουσιάστηκε χθε και μας δείχνουν οι εκθέσεις αυτές ότι σε περιπτώσεις ύφεσης οι προσπάθειες ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να επιβραδυνθούν πλέον και ιδιαίτερα για το 2013 θα πρέπει να μειώσουμε την προσπάθεια αυτή κατά 85 δις αν δεν θέλουμε να έχουμε μια εκρηκτική πλέον αύξηση της ανεργίας. Τρεις ερωτήσεις λοιπόν πιο συγκεκριμένα. Είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε και με άλλους εμπλεκομένους την πολιτική στα πλαίσια των προβλέψεων. Δεύτερον, το θέμα του δημοσίου χρέους προφανώς είναι κρίσιμο και τι σκοπεύετε να κάνετε σε σχέση με το Ταμείο α, α, Απόσβεσης, αν θέλετε. Και τρίτον, η πρωτοβουλία ανάπτυξης και απασχόλησης που ξεκίνησε τον Ιούνιο δεν έχει αποδώσει τίποτα και οι μακροοικονομικές ανισότητες δεν έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ζήτησης και δεν έχουν δημιουργήσει κανένα περιθώριο κίνησης για το σύνολο της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Η Βερόνικα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θετικά εκτιμώ την παρουσία σας ε, ε, και τη δράση σας ως Επιτρόπου και προσδοκώ και ελπίζω ότι θα μπορέσει και ο Επίτροπος Άντορ να συμμετάσχει, κυρίως για τα θέματα της απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να κάνει κανείς ερωτήσεις ε, προς τον Επίτροπο χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς θα αναφερθεί σε σχέση με την απασχόληση αναμένουμε να εξετάσουμε την μελέτη για την ανάπτυξη για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε με τρόπο που πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στις δράσεις. Χωρίς αμφιβολία, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα είναι πάρα πολύ περίπλοκη, πολύ σύνθετη και πιστεύω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τις προτεραιότητες που έχουν, που ξεκίνησαν το προηγούμενο εξάμεινο, αλλά που αδιαμφισβήτα δεν έχουν ακόμα δώσει τα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε και θα ήθελα οι δύο επίτροποι να το σχολιάσουν αυτό, να μας πούν τις απόψεις τους για την κατάσταση ως έχει, τι έγινε μέχρι σήμερα και ποιες προτεραιότητες μπορούν να μας βοηθήσουν να ε, ξεφύγουμε από αυτή την κρίση, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να εξέλθουμε από αυτή την κρίση. Πρώτο σημείο ως προτεραιότητα είναι ο στόχος η στρατηγική Ευρώπη 2020. Η Ευρώπη δεν μπορεί να καθυστερήσει σε σχέση με τη στρατηγική 2020 που πρέπει να οδηγηθεί και να φτάσει σε αυτήν. Πρέπει πρώτα να υλοποιήσουμε τους στόχους μας με σοβαρό τρόπο με αυτά τα οποία δεσμευθήκαμε για τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε με αηφόρο και ευφυή δράση και ανάπτυξη. Έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι πολύ λίγο προχωρήσαμε. Το αντίθετο, μπορεί κανείς να πει ότι οξύθηκε η κρίση περισσότερο. Και πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυξημένα προβλήματα. Λυπούμε για το ότι η αποτελεσματικότητα των πολιτικών προσανατολισμών σε σχέση με το 2012 και η υλοποίησή του ήταν ανεπαρκή όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τη στρατηγική 2020. Είναι αναγκαίο λοιπόν τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τους, ε, τις δεσμεύσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για τις ε, μεταρρυθμίσεις και για την επίτευξη των στόχων αυτών. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας κύριε Επίτροπη. Άλλα θεμελιώδη σημεία είναι η δημιουργία εργασίας και θέσεων απασχόλησης μέσω διαρθρωτικών αλλαγών και μέσω κινήτρων φορολογικών και άλλων για την ανάπτυξη. Είναι αναγκαίο πιστεύουμε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν ευνοϊκά μέτρα για την δημιουργία της απασχόλησης, όπως ε, την μεταρρύθμιση της ε, εργατικής φορολόγησης, ε, της φορολόγησης εργασίας και της φορολόγησης επιχειρήσεων. Είναι θεμελιώδους σημασίας, όπως σε χώρες όπως τη δική μου, να υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Επίσης, κέρια σημασία είναι η σημασία της αγοράς εργασίας που πρέπει να, ολοκλη... να, είναι, ε, να συμπεριλαμβάνει το δυνατόν περισσότερους πολίτες ε, και να μπορέσει η οικονομία έτσι να ενεργοποιηθεί όπως και η ψηφιακή οικονομία. Άλλο από τα κύρια προβλήματα που θα ήθελα να σχολιάσετε κύριε Επίτροπη είναι η ανεργία των νέων η ανεργία των νέων είναι ένα πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Χωρί αμφιβολία στη χώρα μου, στην Ισπανία, είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση από αυτήν που σημειώνεται αλλού. Έχουμε πάνω από 50% των νέων που είναι άνεργοι στη χώρα μου. Γι' αυτό είναι αυτονόητο ότι πιστεύω φυσικά ότι πρέπει να έχουμε μια σαφέστατη στρατηγική για την καταπολέμηση τη ανεργία των νέων. Για το τι πρέπει να γίνει. Τι προτείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, άλλε προτεραιότητε που είναι σημαντικέ είναι μια αγορά πιο προσαρμόσιμη, πιο προσαρμόσιμη πιο ελαστικές δυναμικές για την δημιουργία θέσεων απασχόληση. Δυναμική που πρέπει να αναπτυχθεί. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε πιο δυναμικές λύσεις και επιλογές και πρέπει να σκεφτούμε κυρίως τις γυναίκες τους πιο ευάλωτους τομείς δηλαδή της κοινωνίας μας που πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες και για τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό φυσικά καθώς επίσης και η δημοκρατική νομιμοποίηση Σημαντικό θέμα. Είναι σημαντικό ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και να ακούσουμε, να εισακούσουμε επίση και του κοινωνικού εταίρου και την κοινωνία των πολιτών. Διότι αν πιστεύουμε και θέλουμε, επιθυμούμε οι Ευρωπαίοι πολίτε να μπορούν να υποστηρίξουν μέτρα τα οποία θα λάβουμε, λυπούμε, σα ζητώ να σταματήσετε, έχετε ξεπεράσει το χρόνο. Λοιπόν, λυπούμε γι' αυτό. Αν δώσω το λόγο τώρα στον Επίτροπο Ρεν για το τετράλεπτό του, μόνο τέσσερα λεπτά, ε, να απαντήσει σε ερωτήσεις, κυρίως της Ελίσσα. Μετά θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο, τον υπεύθυνο για θέματα απασχόλησης, ούτως ώστε ταυτόχρονα να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να κάνει και την παρουσίασή του. 12-13 λεπτά δηλαδή. Δεν λέω 14. Διότι κάποιος θα ξεπεράσει το όριο. Λοιπόν, όλοι αν μπορείς να απαντήσεις στον πρώτο γύρο ερωτήσεων και έχεις ε, στη διάθεσή σου 4 λεπτά. Ευχαριστώ Σάρων. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις ερωτήσεις της κυρίας Φερέιρα, θέσατε τρία συγκεκριμένα ερωτήματα κατά πόσον καταρχάς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε την ποιότητα των οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απάντηση είναι ναι. Εξεταζόμαστε σε δημόσιο επίπεδο. Ερευνητικά ιδρύματα αξιολογούν, αναλύουν και επαληθεύουν τις προβλέψεις το ένα το άλλο. Συνεχώς γίνεται αυτή η σύγκριση. Και αν γίνει, οι οικονομικές μας προβλέψεις στέκουν πολύ καλά ε, εν συγκρίση με άλλους διεθνείς φορείς. Είναι συνεχής η προσπάθεια. Και είμαστε πάντα έτοιμοι να βελτιώνουμε τις οικονομικές μας προβλέψεις. Οι επόμενες πλήρεις προβλέψεις για 27 κράτη-μέλη, ανάπτυξη, πληθωρισμός, απασχόληση, όλα αυτά τα στοιχεία που θα αναλυθούν, θα παρουσιαστούν ε, το Φεβρουάριο σαν αποτελέσματα. Μετά, ρωτήσατε για τα, ε, το Ταμείο Διάσωσης και τα Ευρωμόλογα. Θα συμπεριλαμβάνουμε αυτά στο σχέδιό μας και εξετάζουμε εκ του σύνεγγυ στο ζήτημα. Παρουσιάζουμε ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις σχετικά με το πώς αυτό το Ταμείο Διάσωσης Αποπληρωμής και το σύμφωνο μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη να ξεπεράσει τα προβλήματα της μη βιωσιμότητας των δημοσιονομικών και το βάρος των χρεών. Παρομοίως όσον αφορά τα Eurobills θέλουμε να το συζητήσουμε σαν αναλλακτική και να δούμε τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται ούτω ώστε να αποφύγουμε άλλους κινδύνους και να ενισχύσουμε την οικονομική ε, σωστή διαχείριση και να καλύψουμε τον τομέα αυτό των ε, Eurobills. Είναι προφανές ότι αυτά του είδους τα ομόλογα, τα Eurobills, και το Ταμείο Διάσωσης απαιτούν κάποιες αλλαγές της ε, συνθήκης. Και ξέρετε ότι αυτό θα επηρεάσει και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των διαφόρων πρωτοβουλειών, υλοποίησεώς τους. Όσον αφορά την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης, τη σχετική πρωτοβουλία, το ανέφερε κυρία Φοντάνε, το θέμα της ανεργίας, το θέμα της δημιουργίας θέσης απασχόλησης, μεταρρυθμίσεις φορολογικές, πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση. Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις σε πολλές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και άλλες χώρες είναι σημαντικό τμήμα της μεταρρυθμίσεως της οικονομίας και της κοινωνίας. Αφορά τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών και την κοινωνική δικαιοσύνη να αισθανθεί ο λαός ότι λειτουργεί η κοινωνία με δίκιο τρόπο. Με έναν τρόπο που δικαιώνει τον κάθε πολίτη της χώρας. Όσον αφορά την ανεργία, πιστεύω ότι ο Λάσλο θα εστιαστεί από αυτού. Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι χρειάζεται κάτι να κάνουμε. Ανάλογη δράση με την κλίμακα του προβλήματος. Η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 25 εκατομμύρια άνθρωποι και μακροπρόθεσμα αυξάνεται. Αυτό είναι απαράδεκτο σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπου είναι πιο υψηλή ανεργία και όπου η αγορά εργασίας είναι πιο κατακαιρματισμένη έχουν υιοθετηθεί το τελευταίο 18 μήνο πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ήταν πολύ συχνά επίμαχες, αλλά είναι σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και είναι σημαντικό τα μέτρα να εφαρμοστούν. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αισθανθούν ικανές να δημιουργήσουν μόνιμες θέσεις απασχόλησης για τους Ευρωπαίους, κυρίως τους νέους Ευρωπαίους. Εκείνοι που χάνουν τη δουλειά τους θα πρέπει να μπορούν να τύχουν υποστήριξης, ε, να υπάρχουν υπηρεσίες υποστήριξης, να βοηθήσουν να ξαναβρούν δουλειά και η κινητικότητα των εργαζομένων θα πρέπει να διευκολυνθεί όσον αφορά διάφορες ευέλικτες ρυθμίσεις για την απασχόληση. Είναι ακρογωνίως λίθος αυτός της έρευνας που κάναμε για την ανάπτυξη και ο Λάσλο Άντορ θα εστιαστεί πιο συγκεκριμένα από αυτών των ζητημάτων. Καλώς, θα δώσω το λόγο τώρα στον Επίτροπο Άντορ. Δεν ξέρω, θέλετε να κάνετε γενική παρουσίαση που θα καλύπτει τις διάφορες ερωτήσεις που ακούσατε ή δεν ακούσατε. Εσείς αποφασίζετε, έχετε το λόγο και κάνετε ότι... Ορίστε. Επίτροπε, η τρίτη με ερώτηση δεν απαντήθηκε. Πρωτοβουλία για ανάπτυξη και θέσεων το λαμβάνω υπόψη, αλλά δεν υπήρξε χρονική πειθαρχία και πρέπει να προχωρήσουμε. Ξεπεράσαμε τα όρια, λέει η τριτη με ερωτηση δεν απαντηθηκε πρωτοβουλια για αναπτυξη και το λαμβανω υποψη αλλα δεν υπηρξε χρονικη πειθαρχια και πρεπει να προχωρησουμε ξεπερασαμε τα ορια λεει η προεδρος Ίσως αυτό μπορεί να καλυφθεί το ερώτημα στον επόμενο γύρο των απαντήσεων, το τρίτο ερώτημά σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που έφτασα με καθυστέρηση. Θα ήθελα καταρχάς να κάνω μια σύντομη παρουσίαση των θεμάτων που αφορούν την απασχόληση στα πλαίσια της έρευνας και ίσως έτσι να μπορέσω να απαντήσω και σε κάποιες από τις ερωτήσεις τις οποίες άκουσα να τίθενται μετά την αφήξή μου εδώ. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα δύο αυτά έγγραφα περιγράφουν μια πολύ σοβαρή κατάσταση πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της απασχόλησης και στον τομέα των κοινωνικών συνθήκων θα ήθελα να παρουσιάσω συμπερασματικά την ανάλυση την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους συγκεκριμένους τομείς πριν περάσω στις ε, συστάσεις. Δυστυχώς τον προηγούμενο χρόνο η κρίση απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χειροτερεύσει. Είναι η μόνη μεγάλη περιφέρεια παγκοσμίω όπου συνεχίζει να αυξάνεται η ανεργία κάθε μήνα βλέπουμε να αυξάνει το αριθμό των ανέργων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπε ο Αντιπρόεδρος μιλάμε για πάνω από 25 εκατομμύρια πολίτες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε και λίγο πίσω από αυτούς τους αριθμούς που δίνουν έναν μέσο όρο να δούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορετικότητα θα έλεγα. Δηλαδή οι διαφορές από τη μία χώρα στην άλλη αυξάνονται. Η ανεργία στην Αυστρία είναι 4,4% ενώ στην Ισπανία είναι 26%. Κάποιες χώρες αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση καλά, άλλες αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα λόγω και του δημοσίου χρέους και της δημοσιονομικής τους κατάστασης. Θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η κατάσταση υψηλής ανεργίας προέρχεται εν μέρη μόνο από την λειτουργία, οφείλεται εν μέρη μόνο στη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν κάποια θέματα εκεί σε σχέση με τις ρυθμίσεις της εσωτερικής αγοράς, σε σχέση με την επικοινωνία ανάμεσα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Υπάρχουν αδυναμίες της οικονομίας της εργασίας ε, που έχουν αποδυναμώσει κατά κάποιο τρόπο ε, τις δυνατότητες ανάκαμψης στον τομέα της απασχόλησης. Τα βασικά προβλήματα όμως και η αύξηση της ανεργίας είναι καρπός βασικά χαμηλής ζήτησης. Είναι ε, καρπός χαμηλών επενδύσεων λόγω της κρίσης στην Ευρωζώνη και ενός γενικότερα πτωχού θα έλεγα επιχειρηματικού κλίματος σε πάρα πολλές χώρες. Θα πρέπει η αγορά εργασίας να είναι όσο πιο ανθεκτική γίνεται και δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει επίσης την ανάκαμψη. Αυτό ήταν και στόχος του πακέτου που υιοθετήθηκε για την ανεργία τον προηγούμενο Απρίλιο. Οι προτάσεις τις οποίες ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάσταση και να υπάρξει ένα τέρμα στην κατάσταση την αρνητική στον τομέα της απασχόλησης. Η αντιμετώπιση της ε, ανεργίας είναι βασική προτεραιότητα φυσικά ε, και στη νέα έρευνα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάνει λεπτομερείς συστάσεις προς τα κράτη-μέλη στους τομείς αυτούς. Ίσως να υπογραμμίσω κάποια επιμέρους στοιχεία εδώ ε, σχετικά με τις αποφάσεις που πήραμε σήμερα. Πρώτον, χρειάζεται να τονώσουμε την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη ζήτηση για απασχόληση. Η φορολόγηση της απασχόλησης εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ υψηλή, ιδιαίτερα στα χαμηλά εισοδήματα, στους χαμηλούς μισθούς. Και υπάρχουν και ε, επιπλέον επιβαρύνσεις. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις δημιουργικές ε, στον τομέα της απασχόλησης δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας απέναντι σε διακυμάνσεις στον τομέα της οικονομίας και μέσω μεταρρυθμίσεων της ίδιας της αγοράς και μέσω του κοινωνικού διαλόγου αυξάνοντας την ευελιξία της εργασίας έτσι ώστε η απόλυση εργαζομένων να μην είναι η πρώτη απάντηση στην παραμικρή δυσκολία. Απαιτείται επίσης να απλοποιήσουμε την ομοθεσία στον τομέα της απασχόλησης να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την προστασία της απασχόλησης σε προσωρινά απασχολούμενους, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και επίσης θα πρέπει τα επίπεδα αμοιβών να δημιουργούν ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς να δημιουργούν νεοπτώχους. Θα πρέπει επίσης να συνδέσουμε την εκπαίδευση με τον κόσμο της εργασίας γιατί είναι ένα προβληματικό. Ένα στους πέντε δεν βρίσκουν θέση όταν τελειώσουν τις σπουδές τους εύκολα μετά από σπουδές είτε πανεπιστημιακές είτε επαγγελματικές. Θα πρέπει μέσω δυνατοτήτων μαθητείας να συνδέσουμε αυτά τα δύο επίπεδα. Υπάρχει το πακέτο για την απασχόληση των νέων, υπάρχει η πρόταση για τις εγγυήσει για την απασχόληση των νέων, ε, και την βελτίωση ε, των συμβάσεων για την απασχόλησή τους. Θα πρέπει βέβαια να καταπολεμήσουμε και την μακροπρόθεσμη ανεργία. Ε, από τους 26 εκατομμύρια ανέργους, το 11% είναι άνεργοι για πάνω από ένα χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να τονώσουμε τις επενδύσεις στις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τα θέματα της απασχόλησης. Αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι πιο ισχυρές, πιο αποτελεσματικές, να βοηθούν τις μεμονωμένες διαδικασίες αλλά και ομαδικές προσπάθειες έβρεσης εργασίας και τέλος θα πρέπει να τονώσουμε τις κοινωνικές επενδύσεις και να βελτιώσουμε την κοινωνική προστασία οι επιπτώσεις στα εισοδήματα των πολιτών και τα δίκτυα, αν θέλετε, προστασίας έχουν αποδυναμωθεί λόγω της κρίσης. Σε τα επίπεδα έχουν ε, ε, μειωθεί ε, προστασία σε δύο στα δύο τρίτα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα στις πτωχότερες οικονομικά χώρες. Ε, κάποιες ε, πολιτικές για την καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας είναι απαρότητες. Θα πρέπει να συνδέσουμε την κοινωνική προστασία και την προσπάθεια επανένταξης στον κόσμο της εργασίας. Θα πρέπει να αποτρέψουμε τον αποκλεισμό από τον κόσμο της εργασίας. Αυτό όλο το ονομάζουμε κοινωνικές επενδύσεις. Οι κοινωνικές επενδύσεις δεν είναι κάτι το εύκολο, ιδιαίτερα σε περιόδους δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι απαραίτητες οι κοινωνικές επενδύσεις για να αποφύγουμε περισσότερα προβλήματα στο μέλλον να πω ότι η ετήσια έκθεση είναι ξεκάθαρη όταν αναφέρεται σε μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης διαφοροποιούμενα και κοινωνικά φιλικά και για παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των υπηρεσιών έβρεσης απασχόλησης κτλ. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στο πρόγραμμα εγγυήσεων για την απασχόληση των νέων. Είναι επενδύσεις στον τομέα αυτό, αυτές που έχουν γίνει κρίσιμες και θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί και η λειτουργία των συστημάτων κοινωνικής προστασίας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους ε, θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά και στα πλαίσια του πακέτου κοινωνικών επενδύσεων στις αρχές του 2013. Να πω ότι ορισμένες χώρες έχουν προχωρήσει σε βαθύτατες μεταρρυθμίσεις διαφθορτικές της αγοράς εργασίας ανάλογα με τις ε, συνθήκες και τις συστάσεις για κάθε χώρα. Χρησιμοποιούν και ποσά κοινοτικά προς την κατεύθυνση αυτή και μετά από το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ιδιαίτερα για τους νέους. Απαιτείται όμως μεγαλύτερη δράση από τις κυβερνήσεις και από τους κοινωνικούς εταίρους για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να γίνουν πιο ανθικτικές οι αγορές εργασίας και να βοηθήσουμε τα ευάλωτα μέλη των κοινωνιών μας να σταθούν ξανά μόνοι τους. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε μπήκατε στη συζήτησή μας ουσιαστικά με αυτά τα οποία είπατε. Θα έχετε τη δυνατότητα να ξαναπάρετε το λόγο μετά από τις ε, παρεμβάσεις των σκιωδών εισηγητών. Σε ένα δεύτερο γύρο λοιπόν ερωτήσεων θα ακούσουμε τέσσερις παρεμβάσεις μάλλον. Δύο σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής Απασχόλησης και δύο σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Θα ξεκινήσω με τη σειρά. Δηλαδή, ο κύριος Ζων Πολ Γκοζές, εξ ονόματος της Οικονομικής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. 1,5 λεπτό έχετε κύριε Γκοζές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αυτό με ξανανιώνει. Κύριε Επίτροπη, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που η δουλειά που έκανε το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ελήφθη υπόψη, χρησιμοποιήθηκε, το είπατε επανειλημμένα αυτό. Θα δούμε διαβάζοντας το κείμενο το οποίο μας πείτε σήμερα, αν πράγματι αυτό ισχύει, αλλά δεν έχω λόγο να μη σας εμπιστευτώ. Το Κοινοβούλιο δεν εργάστηκε εν και ενώ, μάταια. Όλοι αναφερθήκατε και οι δύο αναφερθήκατε σε μέτρα που δρομολογούνται για τη βελτίωση της κατάστασης, της οικονομικής καταστάσεως και της απασχόλησης. Ποιος δεν θα συμφωνούσε με αυτή την βούληση. Πιστεύω κανείς, βλέποντας την παρούσα κατάσταση που είναι δύσκολη στις διάφορες χώρες. Το θέμα, το ερώτημα αφορά την αξιοπιστία της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι σήμερα η εικόνα που προβάλλει η Ευρώπη είναι διέρεσης. Διχασμένες χώρες που δεν συμφωνούν ούτε επί προϋπολογισμού, ούτε επί τραπεζικής ενώσεως. Και μπροστά στην κοινή τους γνώμη λέγουν άλλα από αυτά που λέγουν ε, και συμφωνούν στις Βρυξέλλες. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι η βούλησή σας, δεν την αμφισβητώ. Αλλά ποια μέσα έχετε στη διάθεσή σας, ούτω ώστε αυτά τα κείμενα, τα καλογραμμένα, τα ισορροπημένα προϊόντα προβληματισμού να καταλήξουν σε μια πραγματική λύση και σε αντιληπτή αποτελεσματικότητα για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την Επιτροπή Απασχόλησης και για το S&D, για τους συστές, ο κύριος Γκουτιέρες. Πριέδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω, κύριε Πίτροπε, αν έχετε συνειδητοποιήσει για την απουσία, την έλλειψη αξιοπιστίας που έχουν τα λόγια σας. Απουσία αξιοπιστίας στους πολίτες και στο Ευρωκοινοβούλιο. Πιστεύω δεν το έχετε συνειδητοποιήσει. Αν το είχατε συνειδητοποιήσει θα είσαστε πιο αυτοκριτικοί στα όσα είπατε. Και χαίρομαι που είσαστε και οι δύο εδώ παρόντες σήμερα. Διότι η πολιτική που αποφασίζει ο ένας των Επιτρόπων έχει επιρροή στους στόχους ε, και στην πολιτική που αφορούν ε, τα μέτρα του άλλου Επιτρόπου. Η ερωτήση μου πρώτη, ποια είναι τα συμπεράσματα που εσείς συνάγετε όταν δεσμεύεστε για παράδειγμα σε σχέση με το προηγούμενο εξάμεινο ότι εφέτος θα είχαμε 0,4% όμως μειώνεται και δεν αυξάνεται και όταν λέτε ότι θα υπάρξει αύξηση πάνω από 1% και όταν έχουμε ελάχιστη ανάπτυξη. Τι πήγε στραβά, τι δεν πήγε καλά. Γιατί πρέπει να το έχετε συνειδητοποιήσει σε σχέση με τι δεσμεύσει ε, που επομιστήκατε πέρσι ότι κάτι δεν πήγε καλά. Δεύτερον, είσαστε διατεθειμένοι να αλλάξετε ε, την πορεία σε σχέση με τα φορολογικά κίνητρα κτλ. Ότι δηλαδή ένας ε, ένα, ένα σημείο αύξηση ή τέλο πάντων ένας βαθμός περικοπής ε, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις. Π.χ. στο τι συμβαίνει στην Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία ότι δίνουμε μια εικόνα ως Ευρωπαϊκή Ένωση που μας γελιοποιεί για να αντιμετωπιστεί η κρίση όπως πρέπει. Τρίτον, είπατε επίτροπε, σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Δρέν το είπε, ότι βλέπετε θετικές προοπτικές για την πρόσβαση στην απασχόληση. Σας ερωτώ πού, πού βλέπετε να υπάρχει τέτοια θετική προοπτική και αν υπήρχε με τι κοινωνικό κόστος θα υπάρχει πρόσβαση στην απασχόληση, ιδιαίτερα για τους νέους. Τέταρτον, εσείς δεσμεύεστε να ε, υπάρξει δέσμευση σε σχέση με τις κοινωνικές δεσμεύσεις στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης σε σχέση με την απασχόληση για τους νέους ε, που είχατε δεσμευτεί και δεν υπήρξε ούτε ένα ευρώ που να δόθηκε σε αυτά. Ευχαριστώ. <laughs> Κακής. Ο κύριος Σκυλακάκης της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής για τους φιλελευθέρους και μετά η κυρία Μάρκεν, Επιτροπή Πασχάλης. Κύριος Σκυλακάκης. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Επίτροποι, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Γνωρίζετε, υπάρχει μια αρχαία ελληνική λέξη, euphemism, εφημισμός, στα αγγλικά euphemism. Μπορούμε να αποκαλέσουμε την πολιτική για την απασχόληση εφημισμό, διότι είναι κατεφημισμόν πολιτική απασχόλησης. Διότι έχουμε ουσιαστικά στην Ευρώπη μια πολιτική ανεργίας και όχι απασχόλησης. Η πραγματική ερώτηση για μένα είναι, για όλες αυτές τις χώρες που έχουμε 25 15-16% ε, ανεργία και όπου έχουμε αργό μη εργαζόμενο δυναμικό προσωπικό πολίτες, σε εκατομμύρια πολίτες άνεργοι. Αισθάνεστε ότι έχετε τα εργαλεία, τα μέσα και εσείς και τα κράτη-μέλη που εμπλέκονται για να κάνετε κάτι πραγματικά, για να καταπολεμηθεί η ανεργία κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Τι λέτε. Merci. Σας ευχαριστώ, Μάρια Νάρκιν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους. Κοίταξα τα ανακοινωθέν τύπου. Και ο κύριος Μπαρόσο είπε ότι βλέπουμε, θέλουμε και οι δύο εξετάζουμε, θέλουμε το, να υπάρξει φιλική οικονομική Εξυγίανση. Ο ορισμό τη τρέλα είναι όταν κανεί κάνει τα ίδια πάντα και περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα. Αυξάνουν οι αποκλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφορέ. Πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι. Πράγματι, χρειαζόμαστε οικονομική εξυγίανση. Ο ρυθμό όμω αυτή τη εξυγίανση, κανεί δεν αμφισβητεί το ρυθμό. Το φάρμακο τελικά θα δηλητηριάσει κάποιου ασθενεί τουλάχιστον και θα μολύνει του υπόλοιπου. Οποιαδήποτε σχόλια κάνω χρωματίζονται από την καταγωγή μου, την Ιρλανδική, που φαίνεται ότι είναι το υθετημένο παιδί της ε, οικονομικής εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής και καμιά φορά αναφέρονται ε, όπως το ΑΕΠ. Πέρσι είχαμε ανάπτυξη 1%, αλλά η διαφορά μεταξύ ΑΕΠ, ε, καθαρίστου εγχωρίου προϊόντο και καθαρού προϊόντο είναι 20%. Το, GN, το ΑΕΠ πέρσι ήταν 7%. Ε, αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να προβληθούν, διότι δεν μπορούμε να θεωρηθούμε ότι είμαστε η επιτυχία ενός μέτρου που δεν λειτουργεί. Η Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί με την εντολή που διαθέτει. Συμφωνώ και πολλέ πολιτικέ σα τελικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα δώσουν αποτελέσματα, έχουν τις δυνατότητες, αλλά βραχυπρόθεσμα. Ε, τι πρόκειται να κάνουμε και τι θα κάνουμε για τους ρυθμούς που ακολουθούνται. Τι ερωτήσει. Το βάρος του χρέους. Άλλαγα ότι είχα 1,5 λεπτό. 10 δευτερόλεπτα λοιπόν τα δημοσιονομικά ε, πώς θα σταθεροποιήσουν το χρέος. Και είναι υψηλότερο το βάρος του χρέους. Όταν είναι υψηλότερο πώς θα κινηθείτε. Θα επανεξετάσετε αυτό το ρυθμό της εξυγίανσης. Και όλες οι ενδείξεις είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους του 2020. Ε, και ποιες είναι οι λύσεις που προτείνετε γι' αυτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξανακούσουμε τους επιτρόπους για να δώσουν απαντήσεις. Πρώτα Επίτροπος Ρεν, μετά Επίτροπος Άντορ και μετά θα ακολουθήσει ο επόμενος γύρος ε, ερωτήσεων. Ε, Επίτροπε Ρεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα του κυρίου Γκοζές σχετικά με την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας όσον αφορά την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ευρωζώνης. Δηλαδή, σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσεως. Όμως, όπως και στη ζωή, και εδώ δεν έχουμε μαύρο, άσπρο. Έχουμε διαφορετικές αποχρώσεις του Θεού ή άλλου χρώματος. Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε αρκετές πολιτικές το τελευταίο εξάμεινο, το καλοκαίρι και μετά. Σε κάποια άλλα ζητήματα όμως το έργο μας έκρεμει και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Παραδείγματος χάρη. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθεροποίησης, ο μόνιμος μηχανισμός, έγινε λειτουργικός τον Οκτώβριο. Είναι το μεγαλύτερο τείχος στον κόσμο, το οικονομικό τείχος προστασίας και δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τα αποτελέσματα. Παρομοίω, έλαβε πολύ σημαντικέ αποφάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τι οικονομικέ ε, συναλλαγέ, ορίζοντα το πλαίσιο και του όρου για ενδεχόμενε παρεμβάσει ε, τη δευτερογενού αγορά. Αυτό είναι κάτι που ηρέμησε τις αγορές και αυτό θα φανεί με χρονική υστέρηση όσον αφορά τη δημιουργία εμπιστοσύνη στην πραγματική οικονομία στην Ευρώπη. Θα θυμόσαστε ότι οι αρχές του χρόνου, περίπου τον Απρίλιο, είχαμε μια αρνητική κάμπη, αν θέλετε. Το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν θετικές εξελίξεις. Είχαμε ανάπτυξη και είδαμε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία ανέκαμπτε. Μετά είχαμε νέες εκλογές, δύο εκλογές στην Ελλάδα, στην Ισπανία. Οι τράπεζες αντιμετώπισαν σοβαρότερες δυσκολίες και δεν ήταν επιστική αντιμετώπιση στην Ευρωζώνη. Με χρονική στέρηση είδαμε μείωση της ανάπτυξης και εξακολουθούμε να υποφέρουμε από αυτό. Όμως, ταυτόχρονα, αναλαμβάνουμε αποφασιστική πολιτική δράση, ούτως ώστε να επιστρέψουμε στην ανάκαμψη. Η απόφαση της Δευτέρας ή της Τρίτης το πρωί όσον αφορά το νέο πακέτο για την Ελλάδα για τη μείωση του βάρους τους χρέους που δεν ήταν βιώσιμο ε, ήταν σημαντική καμπή. Αυτή η απόφαση δείχνει ότι η Ευρωζώνη είναι σοβαρή. Όταν λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να εξασφαλίσουμε την αμετάκλητη πορεία και βιωσιμότητα προς το ευρώ, το εννοούμε. κάποιοι παρατηρητές και κάποιες δυνάμεις της αγοράς είπαν ότι έχουν μείνει πίσω αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στην Ευρώπη. Οι κερδοσκόποι και στοιχηματίζουν στην κατάρρευση του ευρώ και των τραπεζών έχουν μείνει πίσω αυτοί. Είναι η σειρά τους. Όσον αφορά την έξοδο της Ελλάδας. Λοιπόν, Είμαστε σοβαροί για τη βιωσιμότητα του ευρώ και για τη μείωση του χρέους, του βάρους του χρέους της Ελλάδας, ούτως ώστε να είναι βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας και να επιστρέψει στην οικονομική ανάπτυξη και στην ανάκαμψη Ελλάδα. Έγιναν πολλά, αλλά πράγματι πολλά απομένουν να γίνουν και γι' αυτό αυτή η ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω δράση και το, το σημερινό σχέδιο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εμβάθυνση και πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση ε, διευκολύνει τέτοιου είδους ε, δράσεις. Ο κύριος Γκουτιέρες Πιέτο ε, είπε ότι φέτος η ανάπτυξη ήταν μεγαλύτερη από αυτό που προβλεπόταν. Σας εξήγησα, λιγότερη ανάπτυξη, συγγνώμη. Εξήγησα γιατί, διότι απέτυχαν κάποιες πολιτικές πιο πριν, στις αρχές του έτους. Αλλά εν μέρει αυτό οφείλεται και σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στο εξωτερικό περιβάλλον. Και οι δύο παράγοντες είχαν αρνητική συνέπεια όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη φέτος και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, να διορθωθούν αυτές οι αποτυχίες. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να βελτιώσεις επιδόσεις και στα κράτη-μέλη ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Και έτσι θα διευκολυνθεί η επιστροφή στην ανάπτυξη και στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη. Κύριο Σκυλακάκης, τελείωσε ο χρόνος σας λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ και το ερώτημα της Ελίζας αν μπορούσατε να απαντήσετε αυτό που δεν απαντήθηκε πριν. Όσον αφορά το σύμφωνο για την ανάπτυξη και για τις τις χώρες που έχουν πλεόνασμα. Όσον αφορά αυτό το θέμα, ε, τι πλανασματικέ χώρε, Θα επανέλθουμε σε αυτό σε μία-δύο εβδομάδες. Ε, ε, ολοκληρώνεται η έκθεση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να εξισορροπηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Να γίνει αυτό με καλύτερο τρόπο και πιο γρήγορα μέσω μεταρρυθμίσεων στις χώρες τις πλεονασματικές. Πολιτικές που θα διευκολύνουν την εξισορρόπηση της ευρωπαϊκής οικονομίας όχι μόνο με μέτρα στις ελληματικές χώρες, αυτό που συμβαίνει, αλλά και να ληφθούν και μέτρα και στι πλεονασματικέ χώρες. Σχετικά με αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα πράγματα προχωρούν. Στη Γερμανία ο πρόσφατος γύρος διαπραγματεύσεων για τις αμοιβέ οδήγησε σε μέσο όρο αύξηση 5% των αμοιβών στον επόμενο γύρο. Και αυτό υποστηρίζει την εγχώρια ζήτηση και την καλή επίδοση της αγοράς εργασίας στη Γερμανία και το υψηλό επίπεδο απασχόλησης το στηρίζει αυτό στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Αλλά το εξετάζουμε το θέμα και είμαι πολύ πρόθυμος να επανέλθω, να το κουβεντιάσω μαζί σας, να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα της επανεξισορρόπησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Λάσλο Άντορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητά μέλη. Θα ήθελα να διαφωνήσω με αυτούς που λένε ότι η Ευρωπαϊκή κάνει πάντα το ίδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πάντα το ίδιο. Όχι, έχει αλλάξει και στον τομέα της οικονομικής πολιτικής και στα θέματα τα χρηματοοικονομικά. Έχουμε κάνει πολλές προτάσεις, έχουν αναλυθεί πολλές πρωτοβουλίες Πολλές φορές κάποιες προτάσεις δεν έχουν προχωρήσει από το Συμβούλιο βέβαια, αλλά όχι μόνο στο Συμβούλιο. Υπάρχουν επίσης προτάσεις των οποίων η ταχύτητα εφαρμογής καθυστερεί στον τομέα της απασχόλησης. Έχουμε πάρει πολλές νέες πρωτοβουλίες. Αν έχετε προσέξει και γνωρίζω ότι έχετε προσέξει, το πακέτο απασχόλησης του προηγούμενου Απριλίου, Προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε την στρατηγική απασχόλησης και να την καταστήσουμε καταλληλότερη για τις συνθήκες της ε, σοβούσης κρίσης. Αυτό ε, προσπαθούμε να το κάνουμε όχι μόνο επηρεάζοντας ε, τα θέματα της πλευράς της προσφοράς, αλλά προσπαθούμε να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε με πιο αποτελεσματικές δυνατότητες στον τομέα της ζήτησης. Καλύτερα να γίνουν τα πράγματα από ό,τι σήμερα. Προσπαθούμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια ορθότερη διακυβέρνηση της ε, πολιτικής της εργασίας. Είμαστε σε, πολύ, σε συνεχείς και στενός, στενές επαφές με όλους τους ε, εμπλεκομένους έτσι ώστε οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε να ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα στις απόψεις των ε, κοινωνικών εταίρων. σχετικά με τη χρήση του κοινωνικού ταμείου έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο εμείς ε, υιοθετήσαμε σαν Επιτροπή την πρωτοβουλία για τους νέους, ανταποκρινόμενοι στις επιθυμίες των ενδιαφερομένων, βλέποντας ότι αντί για να έχουμε κάποια υφόρο ανάπτυξη, πολλές χώρες γλιστρούν στην ύφεση. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες που επηρεάζουν αρνητικά τη νέα γενιά. Γι' αυτό λοιπόν αναλάβαμε πρωτοβουλίες, αντίθετα από το παρελθόν, πήγαμε στα κρατημέλη που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά προβλήματα, είδαμε ποιες είναι αυτές οι χώρες με τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων και κατά κάποιο τρόπο ανακατευθύναμε τις πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς οι οποίοι με κατεπήγοντα τρόπο αντιμετωπίζουν περισσότερο τις ανάγκες των νέων στον τομέα της εργασίας. Τα ποσά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή φτάνουν περίπου τα 10 δις ευρώ. Δεν αναφέρομαι μόνο στο EFSS αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς την κρίση που συνεχώς βαθαίνει. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, υπάρχει μια νέα πρωτοβουλία όχι μόνο φυσικά το θέμα της πολιτικής για των εγγυήσεων για την απασχόληση των νέων. Ξέρετε ότι αυτό έχει ήδη από το 2010 ενταχθεί στη στρατηγική μας. Αλλά στην αρχή βέβαια όταν είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό υπήρξε μια κάποια χαλαρότητα. Συζητούσαμε γενικά για νέα μέσα έτσι ώστε να <clears throat> τονώσουμε την απασχόληση. Πριν ένα χρόνο όμως, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ε, για την εργασία των νέων, για την απασχόληση των νέων, επανήλθαμε στο θέμα, το ορίσαμε σωστότερα, ε, διαμορφώθηκε ένα πιο ευνοϊκό κλίμα εκ των πραγμάτων και στο Συμβούλιο και ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να καταλήξουμε ε, σε ένα πολύ συγκεκριμένο πακέτο για την απασχόληση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι επαφές μας και με την Ιρλανδική Προεδρία μας δείχνουν ότι οι συζητήσεις στο Συμβούλιο θα πρέπει να είναι ταχύτατες <clears throat> και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθούν το ταχύτερο δυνατόν. Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ στη σημασία των χρηματοδοτικών μέσων. Είναι κομβικά βέβαια για το 2012 και πέραν του 2012 και γι' αυτό είναι λυπηρό θα έλεγα. <clears throat> Επαναλαμβάνω είναι λυπηρό να βλέπει κανείς το πώς εξελίχθηκε η κατάσταση, πώς δεν εξελίχθηκε καλύτερα η κατάσταση στα πλαίσια των συζητήσεων για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 12. Έχουμε ένα κενό χρηματοδότησης και απαιτούνται κάποιες πιστώσεις για να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης των νέων. Ευχαριστώ λέει η κυρία Μπερές. Φτάνουμε τώρα στον τρίτο γύρο ερωτήσεων. Τούρουνεν από πλευρά των Πρασίνων και για τις δύο επιτροπές και μετά ο κύριος Χουντής. Ναι, είμαι η μόνη εδώ που είναι μέλος και των δύο επιτροπών και θα προσπαθήσω να καλύψω και τις απόψεις των πρασίνων από πλευρά. μου. Πρώτα, πρώτα λέτε ότι υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης ε, στο δημοσίο μας τον τύπο. Αλλά υπάρχουν και πολύ αρνητικά σε σχέση με τις προβλέψεις που πρέπει να το αναγνωρίσετε σε πολύ ε, σημαντικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βλέπουμε πολύ χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης για φέτος και του χρόνου. Αύξηση, συνεχιζόμενη αύξηση ανεργίας το 2013 και το 2014. Νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το στοιχείο. Και τρίτον, και πέρσι και φέτος είδαμε αυξημένο χρέος πολλαπλά έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ των έξω να αναγνωρίσει αυτά τα στοιχεία που έχουν σημασία κλειδίου και σε βαθύτερο επίπεδο. Και ερώτηση προς τον κύριο Ρεν πρώτα. Για το μηχανισμό ε, προειδοποίησης ε, είδα ότι προσθέσατε έναν δείκτη στον χρηματοοικονομικό τομέα. Είχε προβλεφθεί όμως στην έκθεση 1176-2011 ότι θα διαδραματίζει το Κοινοβούλιο ένα ρόλο όταν πρόκειται για επικαιροποίηση αυτών των θεμάτων. Ποιο ρόλο μπορείτε να δείτε ότι θα έχει η επικαιροποίηση το Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν. Δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε ότι θα υπάρξει μια μελέτη για την ε, αλληλεξάρτηση σε σχέση με το έλλειμμα και το χρέος στην ε, ζώνη ευρώ. Ίσως ε, δεν το άκουσα αλλά Μπορείτε να μου πείτε τι θα συμβεί, τι προγραμματίζεται και πώς θα χρηματοδοτηθεί η ανταγωνιστικότητα, το μέσο ανταγωνιστικότητας. Και εδώ είναι σημαντικό. Λέτε, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ διότι συμπεριλάβατε την εγγύηση για τους νέους. Είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή Απασχόλησης αυτό. Δεύτερον, για τους πιο ευάλωτους τα μέτρα, είπατε, απλούστευση της νομοθεσίας για την απασχόληση και πιο ελαστικές διεργασίες και ρυθμίσεις για την απασχόληση. Πώς αυτά θα βοηθήσουν τους πιο ευάλωτους, είναι συγκεκριμένη ερώτηση. Ο κύριος Χουντής παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αναφέρομαι στον κύριο Ρεν. Κατά την αρχή της ομιλίας του είπε ότι προσπάθησε αυτή τη βδομάδα να συνδυάσει το ρόλο του αρχιτέκτονα και του πυροσβέστη. Η ερώτηση έχει σχέση με το ρόλο του ως πυροσβέστη στη φωτιά της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Κύριε Ρεν, στην τελευταία απόφαση του Eurogroup σχετικά με το ελληνικό χρέος αναφέρεται σαν προϋπόθεση για να εκταμιευθεί η δόση ότι μέσα στο Δεκέμβρη πρέπει να γίνει επαναγορά ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τη δευτερογενή αγορά και σε τιμές αγοράς 23 Νοεμβρίου. Είναι φανερό ότι αυτοί που θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία θα είναι οι ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία, διότι αλλιώς κατά την εκτίμηση των αναλυτών το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Ωστόσο, κύριε Επίτροπε, δεν έχει αποσαφινιστεί από πού θα βρεθούν αυτά τα κεφάλαια για να γίνει η επαναγορά των ομολόγων. Μήπως θα υπάρξει νέο δάνειο από τον EFSF, θα υπάρξουν έντοκα ομο... γραμμάτια και ακόμα, επειδή αυτό το πρόγραμμα εμφανίζεται ως εθελοντικό, Πώς νομίζετε ότι θα πιστούν οι ελληνικές τράπεζες να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, καθώς οι ίδιες λένε ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον, δεν έχουν κανένα κίνητρο. Άλλωστε υπάρχει και το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών των ελληνικών και αν έχει ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα και ο καταμερισμός. Και τέλος υπάρχει το θέμα με τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο προηγούμενο κούρεμα υποχρεωτικά από την Τράπεζα της Ελλάδας έχασαν πολλά κεφάλαια. Αυτή την περίοδο που δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες θα ακολουθεί η ίδια υποχρεωτική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσα κυρία Πρόεδρε. Θα ακούσουμε τους δύο τελευταίους ομιλητές για να επιτρέψουμε στους επιτρόπους να απαντήσουν σε όλα αυτά που έχουν εγγραφεί. Ο κύριος Πουπάκης και μετά η κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της ανάπτυξης όπως είπατε αποτελεί κορυφαίο ζήτημα γιατί συνδέεται με την προοπτική της ΕΕ αλλά και με την επιβίωση των κοινωνιών όταν μάλιστα ορισμένα κράτη-μέλη με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα όπω η Ελλάδα, η ανταγωνιστικότητα αναζητήθηκε σχεδόν αποκλειστικά μέσα από την συρρήκνωση του εργασιακού κόστου και την περικοπή κοινωνικών δικαιωμάτων, ανακυκλώνοντα, όπω είπατε, την ύφεση, την ενεργεία και επώδυνε κοινωνικέ επιπτώσει. Ποιοι λοιπόν μπορούν να είναι οι βασικοί άξονε του νέου αναπτυξιακού σχεδίου, ώστε η Ένωση να επιστρέψει στην ανάπτυξη χωρί να υπονομεύεται η κοινωνική διάσταση που είναι αναγκαία, αλλά και να προσελκύονται ταυτόχρονα επενδύσεις, χωρίς να δημιουργείται μια Ευρώπη δύο ή και περισσότερων ταχυτήτων. Ευχαριστώ. σα Σας ευχαριστώ η κυρία Άννη Ποδηματά και μετά η κυρία Κράτσα. Κυρία Ποδηματά. Κύριε Επίτροπε, εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ε, ισχυρή απρόσμενη αλλά πολύ επικοδομητική παρέμβαση που κάνατε την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, απευθύνοντα έκκληση λίγε ημέρες, λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup στους εμπλεκό, σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν επικοδομητικό πνεύμα και να υπερβούν την καταστροφική λογική των κόκκινων γραμμών. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω επειδή κάνατε αυτήν την ε, παρέμβαση εξ ονόματος της Επιτροπής και να σημειώσω ότι σε γενικές γραμμές αυτό είναι και το πνεύμα, πιστεύω, της απόφασης του Eurogroup σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματο υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Ε, η μία είναι ε, η δοκιμασία, το εγχείρημα της επαναγοράς χρέους να πάει καλά και θέλω απλώς να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε σίγουρος ότι αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί όπως πρέπει. Και το δεύτερο, κύριε Επίτροπε, επειδή ο πιο ασφαλής τρόπος για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα οποιοδήποτε χρέους είναι η ανάκαμψη και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης και επειδή αυτό είναι και μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του ετήσιου προγράμματος ανάπτυξης που συζητάμε σήμερα. Ε, ωστόσο, οι χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής υποφέρουν από πολύ βαθιά ύφεση. Θέλω να ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε ότι, ώστε αυτό που αναφέρουμε ως βασική προϋόθεση, φιλική προς την ανάπτυξη, δημοσιονομική προσαρμογή, να ισχύσει και για τις χώρες που σήμερα εφαρμόζουν προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κράτσα, μετά ο κύριος Θέρκας, παρακαλώ. Ε, κύριε Επίτροπη, θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς στο θέμα της ανεργίας. Ε, είναι περιττό να τονίσω το πόσο είναι σοβαρό θέμα για τα, το όραμά μας το ευρωπαϊκό και για το πολιτικό, την επιβίωση του πολιτικού μας σχεδίου. Ε, ήθελα να ρωτήσω οι ομάδες δράσης που έχουν συγκροτηθεί στις ε, χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα και θα ε, είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν προγράμματα από τα 82 δισεκατομμύρια ευρώ τα διάθετα, μεταξύ των οποίων και η χώρα μου η Ελλάδα, πώς προχωρούν. Δεν έχουμε νέα καθόλου από αυτή την υπόθεση. Έχετε ήδη αποτελέσματα, υπάρχουν εφαρμογές προγραμμάτων. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας γιατί πράγματι είναι μια επιπλέον πρωτοβουλία που πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Δεύτερον, για το ε, ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ήθελα να ρωτήσω πόσο λαμβάνετε, λαμβάνετε υπόψη στα αξιολόγησή σας και στις συστάσεις κατά κράτος το spillover, ας πούμε η αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνικών οικονομιών. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ επικεντρωμένες οι συστάσεις στο πλαίσιο του κράτους μέλους, ενώ βλέπουμε την αλληλοεξάρτηση σήμερα και τις απρόσμενες συνέπειες που έχει ε, μια οικονομία σε άλλες οικονομίες της ε, Ένωσης και κυρίως της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλεχάνδρο Θέρκας, κύριε Επίτροπη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω, σε ένα τόνο χαμηλόφωνο, να σας πω ότι είμαι πολύ ανήσυχος. Ανησυχώ ιδιαίτερα διότι διάβασα τουλάχιστον την περίληψη αυτού του εγγράφου και βλέπω ότι το συλλογικό σώμα των επιτρόπων δεν άκουσε τίποτα απολύτως από αυτά που έλεγε και είπε το Ευρωκοινοβούλιο επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών και ιδιαίτερα στην έκθεση Τάισεν όταν μιλούμε για την, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Δεν ξέρω αν η περίληψη αυτή φταίει αυτής της, ε, αυτού του εγγράφου. Αλλά αν συμβαίνει αυτό, κύριε Ρεν, ούτε μια λέξη δεν υπάρχει για τη στρατηγική 2020. Συνεχίζεται η ανάλυση ότι το μόνο πρόβλημα, λέει, είναι οι μη ισόρροπες σχέσεις μακροοικονομικά. Και ούτε μια λέξη δεν υπάρχει αυτοκριτικής ε, για την αποτυχία, τις αποτυχίες αυτών των πολιτικών και την ανυπαξία πολιτικής ανάπτυξης. Ούτε μια λέξη για τον κοινωνικό πυλώνα. Το αντίθετο, εξακολουθεί να υπάρχει υπό τον κύριο Φαν απόλυτη απουσία για το ανθρώπινο δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που γίνεται όλο και δυσμενέστερη θέση του που είναι το μόνο δυνατό σημείο για μας να ανταγωνιστούμε στο μέλλον. Μακροπρόθεσμα λοιπόν, ούτε μια λέξη για τους νέους, ούτε μια λέξη για την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Ελπίζω, Επίτροπε, ότι όλα αυτά είναι απλά κάτι που παραμελήσατε, κάτι που δεν το κάνατε, το αμελήσατε σε σχέση και με το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, γιατί ο μόνος τρόπος να αλλάξει η κατάσταση είναι το κοφό Συμβούλιο να ακούσει τη φωνή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβούλιο που ομόφωνα ομιλούν. Και παρακαλώ, να εύχομαι να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Merci. Ε, ευχαριστώ. Θα αντιστρέψουμε τη σειρά. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Άντορ να απαντήσει σε 7 ερωτήσεις, σε 7 λεπτά. Ε, ε, εν συνεχεία ο Επίτροπος Ρεν θα συνεχίσει. Ε, Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό το ότι παραμελήσαμε. Γι' αυτό εμείναμε και επιμείναμε ότι στο MFF θα πρέπει να υπάρξει ένα στεναρό, ενισχυμένο ρόλο ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για του στόχους επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό ακριβώ. Είναι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό. Και επ' αυτού εκεί εμένουμε για να υπάρξει η διασύνδεση μεταξύ των χρηματοοικονομικών μέτρων και της στρατηγικής 2020 έτσι λοιπόν να λειτουργήσει ένα, αυτό το μέσο ως ένα μέσο, ως ένα εργαλείο. Αλλά επίσης ε, και για τα άλλα τα οποία γνωρίζετε. Δεν επαναλαμβάνουμε φυσικά κάθε παρατήρηση και κάθε σημείο σε κάθε έγγραφο και σε κάθε αφορμή που δίνεται με τέτοια έγγραφα. Αλλά αυτή είναι η σωστή θέση να γίνει αυτό και το είπαμε. Και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτό και βρισκόμαστε ακόμα στην πορεία και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να είμαστε υπέρ αυτών των μέσων, αυτών των εργαλείων. Φυσικά θα πρέπει να λειτουργήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με μεγαλύτερη ελαστικότητα. Αλλά αυτό ήδη καταδεικνύεται φυσικά πρέπει να πω σε μια περίοδο συγκυρίας κρίσης και επίσης για την υποστήριξη των νέων. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τούρανεν για την υποστήριξη που έδωσε και δίνει για το μέσο εγγύησης ε, των, για τους νέους σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες αυτό. Το θέμα για τους πιο ευάλωτους, το ζήτημα για τους πιο ευάλωτους και πώς μπορεί να βοηθήσει η απλούστευση. Ίσως είναι θέμα ορολογίας εδώ. Εγώ μίλησα για τον κατακαιρματισμό της αγοράς εργασίας, την πόλωση στην αγορά εργασίας όσον αφορά τους όρους και προϋποθέσεις για τους διάφορους τύπους συμβάσεων και γνωρίζετε ότι είμαστε υπέρ του ότι θα έπρεπε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό βελτιώνοντας ακόμα και τους όρους και προϋποθέσεις και την προστασία ακόμα για τους νέους, για τους εργαζόμενους εκείνους που έχουν προσωρινές συμβάσεις απασχόλησης και που για μεγάλη περίοδο στη ζωή τους θα έχουν την ευκαιρία προσωρινά τουλάχιστον μόνο τέτοιες προσωρινές συμβάσει απασχόλησης να έχουν, αν καν βρίσκουν κιόλα εργασία απασχόληση. Αυτό ως όρος απλούστευση, λοιπόν, μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο για να διευκολυνθούν αυτά. Επίσης, ε, το θέμα για την βοήθεια των νέων και σε σχέση με τις βαλτικές χώρες ε, ε, Λιθουανία, Λετωνία, Σλοβακία και για την δυνατότητα να υπάρχει η δράση team, να υπάρξει η δυνατότητα να υπάρξουν ομάδες δράσης υπέρ αυτών των νέων για να μπορέσουμε να δώσουμε 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτές τις χώρες και να επιτευχθούν αυτές οι δράσεις. Με αυτές τις δράσεις περίπου μισό εκατομμύριο νέων μπόρεσαν σε αυτές τις χώρες ε, να κινητοποιηθούν και να υποφεληθούν. Επίσης, ε, παρόμοια δράση ανελήφθη με τα άλλα κράτη-μέλη που, είναι, που προβλέπονται και στο επόμενο, στην επόμενη φάση ως κλίμακα όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ένας παρόμοιος τύπος ε, δηλαδή κατανομής έργου και προσπάθειας παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, τα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς πάντα το ίδιο να κάνει και τα ίδια κονδύλια να δίνει. Πρέπει να υπάρξει χρόνος για αυτά τα προγράμματα να ευδοκιμήσουν και να δώσουν θετικά αποτελέσματα. Αλλά και η χρηματοδότηση και σε σχέση με τα κράτη-μέλη πρέπει να μας κάνει να δούμε τι πρέπει να γίνει κατά την τρέχουσα ε, επόμενη περίοδο, κατά την επόμενη περίοδο. Ο στόχος μου γενικά είναι για τις επόμενες τρεις επισκέψεις μέσα σε μια εβδομάδα, δηλαδή Νότια Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, χώρες που αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα, τα πιο οξυμένα προβλήματα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Επίσης όλοι πιστεύω ότι θα ήθελε να σχολιάσει το θέμα των μισθολογικών προσαρμογών. Αλλά όσον αφορά το ζήτημα της ανάπτυξης, της εξέλιξης των μισθών, της μισθολογικής εξέλιξης, καθορίσαμε μια γενική αρχή των συνδυασμό δηλαδή παραγωγικότητας και δυναμικής προσαρμογής ή διαμόρφωσης των μισθών. Πρέπει να υπάρξει η εξέλιξη, η ε, προσαρμογή αυτή και με οποιαδήποτε τέτοια προσαρμογή, η διόρθωση θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τους κοινοτικού εταίρους, να γίνεται σεβαστό το κοινοτικό κεκτημένο. Βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου συνεργαζόμαστε με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Κατά την τελευταία μου επίσκεψη στην Ελλάδα συνάντησα επίσης και τους κοινωνικούς εταίρους γνωρίζουμε φυσικά τις δικές τους απόψεις, πως εκείνοι προσεγγίζουν και αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση και πάντα συνεργαζόμαστε και με την κυβέρνηση ώστε να αποκατασταθεί η σωστή λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ρεν. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις ερωτήσεις του Ρούνεν. Το πρώτο σας ερώτημα αφορούσε το νέο δίκτυ του χρηματοδοτικού τομέα στον όλο μηχανισμό της έκθεσης συζητήσαμε με το Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη οργανική Συμφωνία και έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Σούλτς, τον Μάρτιν Σούλτς και στην επιστολή αυτή ενημέρωνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περί του δίκτου που αφορά την οικονομική αυτή σταθερότητα τη χρηματοοικονομική σταθερότητα που είναι ο ενδέκατος δείκτης στην έκθεση. Όσον αφορά το μηχανισμό κατανομής. Μετά τις, το συσχετισμό μεταξύ χωρών πλεονασματικών και λιματικών παραπέμπω στην προηγούμενη μου απάντηση προς την κυρία Φερέρα. Η έκθεση μου για τις των πλενοσματικών χωρών και πώς μπορούν να συμβάλλουν στην επανεξισορρόπηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τις επόμενες εβδομάδες. το ερώτημα. Χρηματοδότηση του μέσου σύγκρισης και ανταγωνιστικότητας που προτείνουμε στο σχέδιό μας για πραγματική οικονομική και νοσματική ένωση. Πώς θα πρέπει να γίνεται η χρηματοδότηση Υποθέτουμε ότι καταρχάς πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία επί του ε, πολιτούς αυτού του, του πλαισίου του... και θα είναι θέμα της Ευρωζώνης και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα συμμετάσχουν και θα αποφασίσουν για τον τρόπο χρηματοδότησης του μέσου αυτού. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Χουντή, για την εξαγορά του χρέους στην Ελλάδα. Σωστά είπατε ότι γίνεται μνήα στη δήλωση του Eurogroup στις τιμές που αναμένεται να μην είναι υψηλότερες από αυτές τις Παρασκευής 23 Νοεμβρίου. Νομικά πρέπει να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Νομικά είναι εγχείρημα που αφορά τις ελληνικές αρχές, κυρίως την ελληνική δημοκρατία και τους ιδιώτες επενδυτές. Και από την Ελλάδα εξαρτάται η υλοποίηση του εγχειρήματο. Μπορώ να πω ότι θα υπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση για ενδεχόμενη εξαγορά χρέους και θα γίνουν αναγκαίες επαφές με, την, ε, με τις ελληνικές αρχές. Κυρία Ποδηματά αναφέρθηκε στο εξή. Κατά πόσο αυτή η συμφωνία του Eurogroup θα λειτουργήσει τελικά στην πράξη. Είναι προσεκτικά συντεταγμένη και σαφής η υποχρέωση που ανέλαβαν τα κράτη της Ευρωζώνης να μειώσουν το βάρος του χρέους της Ελλάδας σε δύο φάσεις δυνατών. Στην πρώτη φάση υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις που ανελήφθησαν για τη μείωση του βάρους του χρέους στο 124% το 2020. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει και άλλη δέσμευση από τις χώρες της Ευρωζώνης να εξετάσουν και ενδεχόμενα και άλλα μέτρα και βοήθεια όπως χαμηλότερη συγχρηματοδότηση των διαθωτικών ταμείων ή περαιτέρω μείωση επιτοκίων για την επίτευξη και άλλης αξιόπιστης μείωσης του, ε, του, του, λόγου ε, ελληνικού χρέους προς ΑΕΠ. Υπάρχει σαφέ χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Η πρώτη φάση θα υλοποιηθεί αμέσως τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Συγκεκριμένη υποχρέωση έχει αναλυφθεί γι' αυτό. Μέτρο, μέτρο ξεχωριστά και υπάρχει και άλλη υποχρέωση ταυτόχρονα μέχρι το 2016 να αποφασιστούν αν είναι αναγκαία περαιτέρω μέτρα για να μειωθεί έτσι περαιτέρω το βάρος το, του χρέους. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει θετικότατο αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη της ελληνικής οικονομίας. Ίσως θα δείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει και εδώ μέσω χαμηλότερης στα διεθντικά ταμεία μέσω χαμηλότερης συγχρηματοδότησης. Πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να συνοχιστεί το χαμηλό ποσοστό της συγχρηματοδότησης και στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που έχει σημαντικό αντίκτυπο. 4-5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της περίοδου. 2,5% περίπου του ΑΕΠ που ακόμα και αν ακούγεται μικρό για κάποιους είναι μεγάλο όσον αφορά την βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας. Το όλο πακέτο απαρτίζεται από 5-6 διαφορετικά μέτρα επέκταση ορίμανσης των, ε, των ομολόγων και μείωση των επιτακίων από τα βασικά ιδρύματα που συμμετέχουν, τους φορείς που συμμετέχουν στο πακέτο. Οι επίσημες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν στην συνεδρίαση του Eurogroup στις 13 Δεκεμβρίου με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης εθνικών διαδικασιών και μετά την αναθεώρηση της καταστάσεως του χρέους μέσω της με τη συνεργασία της Ελλάδας. Η κυρία Κράτσα αναφέρθηκε στα spillovers μεταξύ των οικονομιών των κρατώμενων της Ευρωζώνης. Αυτό είναι στη βάση της ετήσιας έκθεσης και γι' αυτό συντάξαμε αυτή την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονάσματα των τρεχόντων λογαριασμών και κάναμε μεταρρυθμίσεις για να πετύχουμε καλύτερη, ομαλότερη επανεξισορρόπηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο κύριος Τσέρκας Αλόνσο αναφέρθηκε στο σχέδιο, στο προσχέδιο, το blueprint αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο συνάδελφός μου Λοάντορ ήδη απάντησε να πω ότι Υπάρχει ενοιολογική διαφορά μεταξύ των δύο ε, εγγράφων που θετήθηκαν σήμερα. Η ετήσια έκθεση ανάπτυξης αφορά συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής και θέματα που αφορούν το έτος 2013, του χρόνου, το επόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την εφαρμογή πολιτικών. Ενώ αυτό το σχέδιο, το blueprint της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης αφορά ανικοδόμηση, επανεξέταση της όλης αρχιτεκτονικής οικονομικής νομισματικής ένωσης. Δεν καλύπτει όλες τις πολιτικές. Δεν υποτίθεται ότι θα έκανε κάτι τέτοιο να καλύπτει όλα τα θέματα των πολιτικών. Καλύπτει τα θεσμικά θεμέλια ε, της Ευρώπης και πώς πρέπει να ενισχυθούν μια τελευταία κουβέντα για να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που δημιουργεί αυτό που ορίζει αυτό το σχέδιο και ισχυρότερη και πραγματική οικονομική νομισματική ένωση χρειαζόμαστε το 2PAC, τη δέσμη των δύο μέτρων, που είναι τα θεμέλια για περαιτέρω πρόοδο, οπότε πιστεύω ότι θα κινηθούμε πάνω σε αυτό για να προχωρήσουμε και να ανοικοδομήσουμε πραγματικά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριοι Επίτροποι, είναι η δεύτερη φορά που συνεδριάζουν οι Επιτροπές μας, η τρίτη φορά μάλλον που συνεδριάζουμε από κοινού. Και ζητώ συγγνώμη κύριε Επίτροπη, αλλά αυτό αποδεικνύει ότι εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνουμε σοβαρά το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και οι δύο έχετε επιμείνει στη μεγάλη σημασία που έχει αυτή η ετήσια έκθεση των ρυθμών ανάπτυξης. Εγώ εκπλήσωμαι γιατί το ανακοινωθέν τύπου, το οποίο έχει δημοσιευθεί, Ξεκινάει κάπως περίεργα. Λέγεται ότι η έκθεση αυτή είναι η εκκίνηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών με το Σύμφωνο Σταθερότητας και τη Στρατηγική 2020. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν μιλάτε όμως στο επόμενο, περνάτε στην επόμενη φάση, δεν κάνετε καμία αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ταυτόχρονα έχετε και το λεγόμενο blueprint στο οποίο αναφερθήκατε και οι δύο και στο οποίο λέγεται ότι εν ολίγης στην ουσία οι πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να ενισχύσουν την κοινοβουλευτική συζήτηση στα πλαίσια του εξαμήνου μέσω και της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση της έκθεσης για την ανάπτυξη, της ετήσιας έκθεσης για την ανάπτυξη. Λοιπόν, εδώ το ένα κομμάτι του εγκεφάλου σας έγραψε την πρώτη σελίδα, το δεύτερο έγραψε τη δεύτερη σελίδα. Εγώ νόμιζα ότι λειτουργείτε συλλογικά. Αν πραγματικά θέλετε τα κράτη-μέλη να πάρουν σοβαρά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, πρέπει να πάρετε σοβαρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παλεύει εδώ και χρόνια έτσι ώστε ο συντονισμός εκ των προτέρων των πολιτικών μας να έχει κάποιο νόημα. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου όταν θα κάνουμε μία συζήτηση για την ευρωπαϊκή οικονομία, για τη διάγνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, έτσι ώστε να πούμε στα κράτη-μέλη τι κατευθύνσεις πρέπει να ακολουθήσουν για να διορθώσουν τα ελλείμματά τους, τότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι σας σύμμαχοι, κύριοι Επίτροποι και ανεξάρτητα από την ποιότητα των λεγόμενων σας, σίγουρα πρέπει να κάνετε παρακαλώ για την επόμενη φορά μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, την οποία θα οργανώσουμε από κοινού στις 28 Ιανουαρίου, θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και γι' αυτό θα πρέπει να την πάρετε πολύ σοβαρά. Επειδή οι συνθήκες δεν δίνουν, αν θα έλεγα, ε, την δυνατότητα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ετήσια έκθεση ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει ε, να βελτιώσετε τις οδηγίες, τις συστάσεις που κάνετε προς τα κράτη-μέλη. Κάποιοι το είπαν σήμερα για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι των εργασιών, εμείς δεν εκπλησόμεθα γιατί αυτή η πορεία την οποία ακολουθούν τα κράτη-μέλη παραμένει η ίδια, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης διορθώνονται προς τα κάτω είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα χθε το ίδιο ακριβώς έκανε και ο ΟΣΑ. Ε, ευχαριστούμε και την Διευμηνία, γενικά λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ και την Συμπρόεδρο και θα συναντηθούμε ε, σε μια αντίστοιχη τέτοια ε, ευκαιρία στις 28 Ιανουαρίου.